So, then I would like... Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην ακρόαση ε, της ε, επιτρόπου Γιούτα Ουρπιλάινεν από τη Φιλανδία, αρμόδια για τις ε, διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Έχουμε τρεις ώρες στη διάθεσή μας, οπότε περάσουμε κατευθείαν στο διάτα αυτά. Καλώς κυρία Γιούτα Ορπιλάινεν, είστε υποψήφια επίτροπος για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτή την ακρόαση. Ξέρουμε πως ε, και εσείς αδειμονείτε όπως και εμείς. Και πριν ξεκινήσω θα ήθελα εν συντομία να σας ε, αναφέρω κάποια διαδικαστικά και το πλαίσιο της δημόσιας ακρόασης. Καταρχήν, με βάση τι κατευθυντήριες γραμμέ για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τον υποψήφιο επίτροπο βάσει των γενικών ικανοτήτων του, την προσήλωσή του στην ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική του ανεξαρτησία. Επίση, αξιολογεί τι γνώσει του κάθε υποψηφίου επιτρόπου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό του και τι ε, ικανότητε επικοινωνία που έχει. Πριν την δημόσια ακρόαση, η κυρία Ουρπιλάινεν απάντησε γραπτός σε ένα ερωτηματολόγιο που της είχαμε στείλει και οι γραπτές απαντήσεις έχουν μοιραστεί και μάλιστα μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες ε, στους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για την διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης. Τώρα, πώς θα διαρθρωθεί η σημερινή συζήτηση η υποψήφια επίτροπος καλείται να προβεί σε μια προφορική ε, εναρτήρια δήλωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Στη συνέχεια θα έχει 5 λεπτά προς το τέλος συνεδρίασης για τα καταληκτικά της σχόλια. Μετά την εισαγωγή θα υπάρξει χρόνος για 25 ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Και μάλιστα η συζήτηση θα γίνει με βάση χρονοθυρίδες πεντάλεπτες, ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση από την υποψήφια επίτροπο. Σε περίπτωση που υπάρχει επερώτηση, ε, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό και η απάντηση το ίδιο, θα είναι μονόλεπτη. Ο πρώτος γύρος ε, επτά ερωτήσεων θα υποβληθεί από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο δεύτερος γύρος θα παρτίζεται από 18 ερωτήσεις βάσει της συνολικής κατανομής των ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και επίσης ε, θα υποβάλει ερώτηση και ένας εκπρόσωπος μη εγγεγραμμένων μελών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρήσετε πιστά το χρόνο που δικαιούστε. Σήμερα Έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες, οπότε όλοι οι ομιλητές δίνονται να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα, αλλά σας θέρμο παρακαλώ να μιλάτε αργά, ώστε να σας προλαβαίνω και οι διερμηνείς και να μεταφέρω σωστά το μήνυμά σας. Επίσης, η συζήτηση μεταδίδεται στην, ζωντανά στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα έχετε πρόσβαση και σε μία ε, σε ένα βίντεο τη ακρόαση στην ίδια στο σελίδα. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στην υποψήφια επίτροπο, θα ήθελα να πω λίγα λόγια ε, επιστώντα την προσοχή σα σε πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μα θέματα, ευελπιστώντα σε πολύ στενή συνεργασία και αγαστή συνεργασία με την υποψήφια Επίτροπο. Καταρχήν, μία από τι σημαντικότερε μεταρρυθμίσει που έχουμε αφορά το Μηχανισμό γειτονία ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία, το NDICI. Ελπίζουμε ότι θα γίνει πιο αποτελεσματικό, θα προβληθεί καλύτερα και θα συμβάλλει στην καλύτερη προβολή της αναπτυξιακής, της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντική ανάπτυξη, ανάμειξη συγγνώμη, και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ο ρόλος ε, της υλοποίησης των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικοποιημένα με ποσοτικοποιημένους στόχους και μέτρα. Ήδη έχει περάσει ένα τρίτο του χρόνου που έχουμε για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και προσβλέπουμε στην άμεση εφαρμογή της στρατηγικής. Επίσης, η συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ μετά το Κοτονού μας ενδιαφέρουν. Έχουμε επιμείνει με δύο ψηφίσματά μας τη συμπερίληψη ε, της ενισχυμένης κοινοβουλευτικής διά, διάταξης με ε, ισχυρότερη διακοινοβουλευτική συνέλευση ΑΚΕ. Επίσης, γνωρίζετε πως, ε, πόσο έντονες είναι οι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για τη συμμετοχή του στην σύναψη και ολοκλήρωση των μελλοντικών συμφωνιών. Και πάλι θερμά καλωσορίζω την υποψήφια επίτροπο και της δίνω το λόγο. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμε Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας ως υποψήφια επίτροπος. Θα ήθελα πρώτα να σας πω δύο λόγια για μένα, για τους στόχους μου και για το πώς πιστεύω ότι μπορούμε από κοινού να τους υλοποιήσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι ουδέποτε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα βρισκόμουν εδώ, σε αυτό το έδρανο, όταν ε, συμμετείχα στην εκστρατεία στην ηλικία των 19 ετών για την ένταξη της Φιλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε μπορούσα να το διανοηθώ, όταν συμμετείχα στις συνεδριάσεις ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ε, ε, Νεολαίας για τα κοινωνικά θέματα. Ούτε όταν συνείδησα και προείδρευσα μιας φιλοευρωπαϊκής οργάνωσης νεολαίας στη Φιλανδία. Ούτε μπορούσα να το φανταστώ όταν πήγα με το πρόγραμμα Έρασμος στη Βιέννη και σπούδασα μουσική μαζί με άλλους Ευρωπαίους. Και τότε ανέπτυξα παρόλα αυτά στα νιάτα μου μια ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και τότε ανέπτυξα την ακράδαντη πεποίθησή μου ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι θετική και για την Ευρώπη, αλλά είναι ευεργετική και για τον κόσμο. Και η ευρωπαϊκή μου ταυτότητα και η πεποίθησή μου στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με καθοδήγησαν στη σταδιοδρομία μου μέχρι σήμερα στον πολιτικό μου βίο ως βουλευτή, Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά με, με ενέπνευσαν και στην προσωπική μου ζωή ως στο, στην κοινωνία των πολιτών και ως ε, ειδική εντεταλμένη για διαμεσολάβηση σε ειρηνευτικά θέματα. Η ευρωπαϊκή ταυτότητά μου και η πεποίθησή μου σε μια όλο και πιο στενότερη και ισχυρή ένωση με έφεραν εδώ μπροστά σας και πιστεύω και ελπίζω ότι με την έγκρισή σας θα γίνω και εγώ μέλος του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να με πιστέψετε. Βρίσκομαι εδώ απέναντί σας <clears throat> με έμπνευση ταυτόχρονα αλλά και ταπεινοφροσύνη γιατί πιστεύω ταπεινά ότι η συμμετοχική αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν πολύ σημαντικές τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο και μας επηρεάζουν. Οι κλιματικές αλλαγές, η ψηφιοποίηση, η μετανάστευση, η κινητικότητα, αλλά και ανισότητες είναι μερικές από τις αλλαγές και τις τάσεις αυτές. Επειδή υπηρέτησα σε οργανώσεις της ε, κοινωνία των πολιτών, αλλά και στο κοινοβουλευτικό έργο για θέματα εξωτερικών ε, ζητημάτων και αναπτυξιακά, ε, είμαι προσιλωμένη στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, στην συνδρομή των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προσφέρθηκα να προεδρεύσω στην, Διεθνή, ε, στην Εθνική Συγγνώμη Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και θεώρησα ιδιαίτερα σημαντικό να ε, φέρω σε συζήτηση διάφορα, διαφορετικά υπουργεία και ενεχομένους, γιατί πιστεύω ότι μόνο με συνεργασία μπορούμε να υλοποιήσουμε σημαντικούς στόχους. Τώρα που η εκλεγμένη πρόεδρος ε, διάλεξε τον ίδιο τρόπο, ε, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί στις επιστολές με τα καθήκοντά μας δηλώνει η κυρία Φοντερ Λάινεν ότι συλλογικά είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και είμαι υπερήφανη για τη σφαιρική προσέγγιση που υιοθετεί και προτίθεμαι να στηρίξω πλήρως αυτή την ε, προσπάθεια και στις εσωτερικές και τις εξωτερικές μας πολιτικές. Είμαι πεπισμένη ότι το θεματολόγιο του 2030 μας δίνει μια χρυσή ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ευρωπαία ε, Επίτροπος για τις διεθνείς εταιρικέ σχέσεις θα πρέπει να υλοποιεί του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. Στόχος μου είναι να εξαλείψουμε τη φτώχεια χάρη στη διεθνή συνεργασία και αναπτυξιακή βοήθεια. Η ευθύνη μας παγκοσμίω φαίνεται και στις συνθήκες και ευθυγραμμίζεται με τι αξίε μα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Δική μου φιλοδοξία είναι να το επιτύχουμε αποτελεσματικά και με στρατηγικό τρόπο και παρακολουθώντας τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια πραγματικότητα. Η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης εξυπηρετεί και τα δικά μας ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γιατί μιλούμε για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Μιλούμε για την ε, ανασφάλεια του κόσμου, για τις συγκρούσεις που εξαναγκάζουν τον κόσμο να εγκαταλείψει τις αιστείες του και να μεταναστεύσει. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν ε, ασχοληθώ με την πολιτική, ήμουν δασκάλα. Η παιδεία, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα που μου είναι πολύ προσφυλές. Ένας ε, βιώσιμος ε, κόσμος χωρίς αποκλεισμού και με ισότητα προϋποθέτει και ισότιμη πρόσβαση των πάντων στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Έχουμε πολλές στάσεις. Ε, η παιδεία λοιπόν μπορεί να, αλλάξει, να, συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας για το κλίμα ή το περιβάλλον. Ο ρόλος της παιδείας είναι τεράστιος στην προετοιμασία των ε, επόμενων αγορών απασχόλησης ε, και την προσαρμογή του στον ψηφιακό κόσμο. Είμαι υπέρ του στόχου του 20% για την ανθρώπινη ανάπτυξη στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι σαφής ο στόχος μου αυτός. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, πιο ευπαθείς περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το ίδιο για παράδειγμα και η βασική εκπαίδευση, η εκπαίδευση της προσχολικής ηλικίας και η εκπαίδευση των νεαρών κοριτσιών. Και τώρα έρχομαι σε ένα πιο προσωπικό ζήτημα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιμόρφωση και η χειραφέτηση των γυναικών, των κοριτσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προαπαιτούμενο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμού. Γνωρίζω τι σημαίνει να σπάει κανεί τις γυάλινε οροφέ, γιατί ήμουν πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματο τη Φιλανδίας και ήμουν και η πρώτη υποψήφια Φιλανδία Επίτροπος. Οπότε θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω για τη βαθύτατη πεποίθησή μου να δώσω προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, προκειμένου να γίνει οριζόντιο θέμα σε όλα τα προγράμματα πολιτική μα. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στην καταπολέμηση της ανισότητας και στην εξάλληψη της φτώχειας. Με ποιο τρόπο όμως θα τα επιτύχουμε όλα αυτά. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε σύγχρονες ε, εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάλογα με τις προτεραιότητές μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τέτοιες πρωτοβουλίες φυσικά απαιτούν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μπορούμε να δείξουμε στους εταίρους μας ότι θέλουμε σοβαρά ε, και υπεύθυνα να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και θα συνεργαστούμε προκειμένου να διευκολύνουμε μια συμφωνία για το Μηχανισμό γειτονία Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. Τη σήμερα ημέρα τα παραδοσιακά μέτρα παρα... χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας δεν αρκούν. Δεν αρκούν για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν αρκούν για να σφυριλατήσουμε τι εταιρικέ σχέσει που θα ανταποκρίνονται στις νέε πραγματικότητες. Ω Ευρωπαίο Επίτροπο, θα σας υπόσχομαι ότι θα χρησιμοποιήσω τη βοήθειά σας για να δημιουργήσω μόχλευση για μεγαλύτερο εθνικό εισόδημα και περισσότερη ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα, του ιδιωτικού κεφαλαίου. Η αναπτυξιακή πολιτική του 21ου αιώνα θα πρέπει να αξιοποιεί όλα τα μέσα και του μηχανισμού για να δημιουργεί περισσότερε επενδύσει, περισσότερε θέσει απασχόληση, καλύτερη νομοθεσία και βελτιωμένη διακυβέρνηση. Αυτό προποθέτει την αξιοποίηση στο έπακρο του εξωτερικού μας επενδυτικού σχεδίου. Ο νέος τίτλος και του χαρτοφυλακίου μου, ε, που είναι πιο σύγχρονος και μιλά για διεθνείς εταιρικέ σχέσεις, ε, μας εστιάζει στην πολυμέρεια και τη συνεργασία μεταξύ ισότιμων εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί από μόνη της ε, να σώσει τον πλανήτη και να προετοιμαστεί για το μέλλον. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία από της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της. Θα πρέπει χέρι με χέρι να προχωρήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θα είναι ο θεματοφύλακας της πολυμέρειας και μιας ε, παγκόσμιας τάξης που θα στηρίζεται σε κανόνες. Η συνδυασμένη ε, ικανότητα βοήθειας ε, των κρατών μελών και των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνεκτικά για να προωθηθούν οι αρχές, οι αξίες και οι στόχοι μας και επιτόπου στις χώρες εταίρους, αλλά και σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το 2015, όταν η παγκόσμια κοινότητα πέρασε από τους στόχους ε, της χιλιετίας, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, εγκατέλειψε την, το διαχωρισμό βορρά-νότου, δωρητή και αποδέκτη, ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου. Η παγκόσμια κοινότητα δημιούργησε μια προοπτική φιλόδοξη ε, με κοινή συμφωνία που θα επωφελεί ε, τους πάντες. Και ως Ευρωπαίοι υποψήφια επίτροπος ε, θα εξασφαλίσω την ευθυγράμμιση και την στεναρή προσπάθεια υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ισχυρές εταιρικές σχέσεις με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία και τον Ειρηνικό μπορούν να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε σε πολλά ζητήματα. Τέτοιες ε, περιεκτικές ε, και συνολικές εταιρικές σχέσεις θα μας επιτρέψουν να απελευθερώσουμε ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως η διαχείριση της μετανάστευσης και όλα αυτά χάρη στη συνεργασία μας. Αν με εγκρίνετε ως Επίτροπο, πρόθεσή μου είναι να αξιοποιήσω την Ευρωαφρικανική Συμμαχία για τις βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης και να τη μετατρέψω σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αφρική. Και στην προσπάθεια μου αυτή θα συνεργαστώ με τον ύπατο εκπρόσωπο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους επιτρόπους. Η εταιρική σχέση με τη γειτονική μας Ήπειρο έχει ε, ενισχυθεί αναβαθμιστεί προ όφελο και των δύο υπήρων, με ανάμειξη και του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω αυτό το δρόμο. Θα πρέπει να βαθύνουμε τα κοινά μας ενδιαφέροντα και την ικανότητα, την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες από κοινού. Ε, το παλιό αφήγημα ότι η Αφρική είναι ασταθής ε, και φτωχή ήπειρος θα πρέπει να εγκαταληφθεί. Θα πρέπει να στρέψουμε τα νότα μας σε αυτή την παροχημένη αντίληψη. Θα πρέπει να ανοίξουμε τις αγκάλες μας προς την Αφρική που είναι μια νέα ήπειρος ε, ε, ελπίδας και ευημερία. Επίσης, προτεραιότητά μου θα είναι να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ μετά το Κοτονού. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μια σύγχρονη στρατηγική και σημαντική συμμαχία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ε, Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού και μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να εξυπηρετεί τα κοινά μας συμφέροντα και τους λαούς όλων των χωρών. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα πιστώ προσπαθειών για να αναδείξω την κατάλληλη κοινοβουλευτική διάσταση αυτής της μελλοντική εταιρική σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντλεί την ισχύ της από τα θεσμικά της όργανα, από όλα τις τα θεσμικά όργανα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω έμφαση στην προσήλωσή μου στη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους θέλουμε να εδραιωθεί ο ηγετικό μας ρόλος στην διεθνή συνεργασία και στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και ως ε, κοινοβουλευτική πιστεύω ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι πολύ σημαντική και θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξάρω αυτή την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την ευαθύνω και να την ενισχύσω. Βρίσκομαι εδώ για να ακούσω τις, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα και τις παρατηρήσεις σας και την εμπειρία σας. Θα συνεργαστώ στενά με τον ύπατο εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να καταστήσουμε την Ευρώπη ένα σημαντικό διεθνή παράγοντα με μεγάλη επιρροή και στο πνεύμα της Γεωπολιτικής Επιτροπής που ανήγγειλε η εκλεγμένη πρόεδρος Ούρσουλα Φοντερ Leyen, προτίθεμαι να συνεργαστώ στενά και με άλλους επιτρόπους που τα χαρτοφυλάκια τους επηρεάζουν τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τα κράτη-μέλη ώστε να αναλύουμε από κοινού, να προγραμματίζουμε από κοινού και να εφαρμόζουμε από κοινού τις πολιτικές μας και να υλοποιήσουμε το στόχο του 0,7 του ακαθάριστου εχώριου εισοδήματο για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ίσως είναι ο σημαντικότερός μας σύμμαχος και θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο, στην καρδιά του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να αναμίξουμε την κοινωνία των πολιτών όσο περισσότερο γίνεται στην διαμόρφωση των πολιτικών και στην ε, σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων μας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόμαστε την πολιτική για τον πλανήτη μας, για την ανθρωπότητα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από εμά να αναλάβουμε δράση. Η νεολαία είναι πιο απαιτητική τα παιδιά μας αξίζουν να βάλουμε τα δυνατά μας. Θέλω να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας και θα πρέπει να εμπνεύσουμε και εμπιστοσύνη στους εταίρους μας ότι είμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη ε, και να καταλάβουν οι πολίτες το σκεπτικό και τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού μας έργου να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη ε, στους πολίτες για τα θεσμικά μας όργανα. Γιατί, αν, ε, γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να έχουμε ένα πιο ισότιμο κόσμο. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας ακούσω και να προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you for uh, that opening statement. Σας ευχαριστούμε για αυτή την αρχική σας ομιλία, υποψήφια επίτροπε, και τώρα θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Χάνμπεν από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κυρία Επιτροπέ, υποψήφια Επιτροπέ. Θα ήθελα να ε, διαβάζω την ερώτησή μου στα ουγγρικά. Ε, σας ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, η μεταναστευτική κρίση του 2015 μας έδειξε ότι στη Μέση Ανατολή και γενικότερα στην Ασία η οικονομική και πολιτική κατάσταση είναι ασταθής και μπορεί να ε, φέρει σε με αστάθεια και να θέσει σε κίνδυνο και τη δική μας σταθερότητα. Οι αδύναμες κυβερνήσεις ουσιαστικά οδηγούν στο να χάνουν ε, και στις χώρες προέλευσης τους οι πολίτες τα δικαιώματά τους. Για τις χώρες αυτές λοιπόν της μετανάστευσης, τα γενεσιουργά αίτια πρέπει να τα ε, καταπολεμήσουμε στην ε, πηγή τους. Θα πρέπει να μπορούν οι άνθρωποι να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους στις χώρες τους, εκεί από που κατάγονται, παρά να διακινδυνεύουν τη ζωή τους προσπαθώντας να μεταναστεύσουν αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ε, βασιστεί σε αυτά τα θεμέλια και να γίνουν και σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Εγώ ίδιος, όπως και η ομάδα μου, ε, το ΕΛΚ, θέλουμε να σας θέσουμε την εξής ερώτηση. Τι σημαίνει για σας το δικαίωμα της Παραμονή. το δικαίωμα της παραμονής ε, κάποιου στη χώρα προέλευση του. Για σας αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των πολιτών στις χώρες τους. Κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ευρωβουλευτά, κύριε Χόλβενη. Ευχαριστώ και εσάς και όλους τους συντονιστές για τις συζητήσεις που είχα μαζί σας πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω όλους τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών δυνάμεων του Κοινοβουλίου. Συζητάτε και ρωτάτε ποια είναι η σχέση μεταξύ αναπτυξιακής πολιτικής και μετανάστευσης. Κατά την άποψή μου, είναι θέμα γενεσιουργών αιτίων. Υπήρξα ειδική ε, εντεταλμένη για τα θέματα ειρήνευσης και μάλιστα έχω ταξιδέψει πολύ στην Αφρική. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ήταν ε, στιγμές δραματικές ε, που σπαράζουν την καρδιά όταν συναντάει κανείς νέους στην Αφρική που έχουν χάσει την ελπίδα για το μέλλον. Όμως το καταλαβαίνω κιόλα. αν δεν έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, αν δεν έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας, στην αγορά εργασίας. Τι πίστη να έχουν στο μέλλον τους. Από αυτήν λοιπόν την πρόπτικη πρέπει να πω το εξή. μέσω της αναπτυξιακής μας συνεργασίας μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης της χώρες προέλευσης και τις ε, χώρες εταίρους μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω των επενδύσεών μας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ούτω καθεξής. Βεβαίως, το συνολικό πλαίσιο για αυτού του είδους τη συνεργασία είναι η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ανέφερα και στην ανακτήρια ομιλία μου. Επερώτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Άρα, όπως σωστά είπατε, αυτό που χρειάζεται στην Αφρική είναι επιτόπου να επέλθουν κάποιες σοβαρέ αλλαγέ. Γι' αυτό λοιπόν σα ζητώ επίμονα πρωτού και εμείς αποφασίσουμε, ε, να μας πείτε αν στην Αφρική, σε άλλες χώρες της Ασίας, είστε σε επαφή με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή πολιτικούς ηθήνοντες από τις χώρες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας που χρησιμοποιεί να έχει και πιο συγκεκριμένους στόχους να αξιοποιήσει και το ε, σκέλος της αναπτυξιακής συνεργασίας και το εργαλείο για την γειτονία. Θα ε, αξιοποιήσετε τα εργαλεία αυτά για να ικανοποιήσετε τους στόχους της αναπτυξιακής ε, πολιτικής. Είμαι πανέτοιμη να οργανώσω διάλογο και με εσά και με όλες τις πολιτικές ομάδες και με όλες τις ομάδες του Κοινοβουλίου και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβανομένων. Ο διάλογος ήταν ε, πηξίδα για τον πολιτικό μου βίο, παρόλο που δεν υπάρχει πάντοτε ταύτιση απόψεων. Πάντως, πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να έχουμε ε, μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική και μελλοντικά είναι να χτυπήσουμε, να ε, παρέμβουμε στο επίπεδο των γενεσιουργών αιτίων. Πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στις χώρες προέλευσης, αλλά και σε άλλες χώρες εταίρους. Είναι ο μόνος τρόπος να φέρουμε ελπίδα στη ζωή των ανθρώπων στις κοινωνίες αυτές. Και είμαι έτοιμη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου στη δουλειά μου ως μέλος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μπούλμαν από τους σοσιαλιστές. Καλώς ήρθατε κυρία υποψήφια επίτροπε εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών στο Κοινοβουλίο. Σωστά λέτε ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι χρυσή ευκαιρία για όλους μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η τελευταία μας ευκαιρία ίσως για να πετύχουμε να καταπολεμήσουμε την ακραία φτώχεια και να αντιμετωπίσουμε σημερινές δυσκολίες όπως τις κλιματικές αλλαγές ή την ε, διόγκωση των ανισοτήτων ή την πολιτική αστάθεια, θα ήθελα να προσθέσω. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να μπούμε και πάλι στο σωστό δρόμο, πώς μπορούμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να έχουμε έναν διεξοδικό δικό χάρτη που προς στιγμή μας λείπει, και σε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο και πώς μπορούμε καλύτερα να παρακολουθούμε και να κάνουμε σωστή κατηγοριοποίηση με δείκτες την επίτευξη των στόχων. Έχουμε δει τα τρία σενάρια της απερχόμενης Επιτροπής και σαφώς προτιμούμε το πρώτο. Είναι το μόνο το οποίο μα ε, επιτρέπει να έχουμε κάποιε ελπίδε για την επίτευξη των στόχων. Είμαστε λοιπόν περίεργοι να μάθουμε κατά δικά σα σχέδια. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για αυτή την τόσο κέρια ερώτηση. Καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αυτό το θέμα ήταν πάντοτε για μένα προτεραιότητα. Όταν ήμουν υπουργό Οικονομικών, θεωρούσα πολύ σημαντικό να κοιτάξω το σκέλος και το, το επίπεδο των ανισοτήτων. Πιστεύω όμω ότι οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη και η ατζέντα του 2030 είναι κάτι σαν πηξίδα για μένα. Θα έπρεπε να είναι αυτό που με οδηγεί εμένα και όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί στη δουλειά μα. Δεν πιστεύω, δεν καταλαβαίνω πώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη μόνον μέσω αναπτυξιακή πολιτική. Πρέπει να έχουμε μια σφαιρική στρατηγική για να τους επιδιώξουμε. Γι' αυτό χάρηκα τόσο πολύ που η υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ρητός σε πολλές επιστολές αρμοδιοτήτων ότι όλο το κολέγιο των επιτρόπων θα είναι ε, συνυπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα εργαλείο που έχει αναφέρει μεταξύ άλλων είναι ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, και εγώ είμαι πέρα αυτής της ιδέας, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο για την υλοποίηση των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας, ίσως. Αλλά όπως είπα στην ανακτήρια ομιλία μας, πρέπει να υποστηρίξουμε και τις ε, χώρε Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουν τι δικέ του ε, ε, εθνικές και περιφερειακού επίπεδου στρατηγικέ για την επίτευξη των στόχων. Διότι Το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να είναι κοινό, αμοιβαίο. Δεν μπορεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να το επιδιώκει και να το υλοποιεί. Πρέπει όλη η κοινωνία του πλανήτη να ασχοληθεί με την επίτευξη. Επερώτηση. Ε, και στην εναρτή ομιλία σας είπατε ότι δεν πρέπει να φέρνουμε σαν τη διαστολή το βορρά με τον νότο αλλά την ε, ιδέα πιο πολύ ότι όλοι είμαστε χώρε σε κατάσταση ανάπτυξης και όλοι έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αναφέρατε το εξάμεινο. Τι σημαίνει αυτό για το χαρτοφυλάκιό σα, διότι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το περιθωριακό για τη δουλειά σας, το δευτερεύον, αλλά είναι πρώτη τη σημασία για το τι θα αναλάβετε. Οι χώρε μα λοιπόν από όλε τι περιοχέ συνεργασία του κόσμου ε, θα έχουν ε, κάτι να συνεισφέρουν εδώ. Ποια είναι η εντύπωσή σα λοιπόν, πώ μπορούμε να οργανώσουμε τα εσωτερικά, τι εσωτερικέ υποθέσει τη Ευρώπη, τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, την εμπορική μας πολιτική, μέσα από την ε, οπτική γωνία, την προπτική των εταίρων μας, με τους οποίους θα πρέπει να πετύχουμε στόχους ενός κοινού δικού χάρτη. Κυρία Επίτροπε, ως προς τις αρμοδιότητές μου και τις εταιρικέ σχέσεις. Νομίζω ότι αυτή η αρμοδιότητα το διεθνείς εταιρικέ σχέσεις έχει καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Όπως είπατε κι εσείς ο ίδιος, αποστέλει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα προς τις χώρες εταίρους. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την απλοϊκή σχέση ε, χορηγού δωρητή. Θέλουμε ισότιμες εταιρικές σχέσεις. Όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο δεν μπορούν από μόνοι τους να καταφέρουν κάτι. Πρέπει τα κράτη-μέλη να εμπλακούν, να λάβουν δράση στην όλη διαδικασία. Και από είπα προηγουμένως, νομίζω το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό νέο εργαλείο για να επιδιώξουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Σαλτ από τη Ρινιού, επόμενος Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Άκουσα με μεγάλη χαρά τα εισαγωγικά σας σχόλια. Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα που περνάει μέσα από το δικό σας χαρτοφυλάκιο, γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος ε, παίκτη στην αναπτυξιακή βοήθεια παγκοσμίω. Ισοτιμία λοιπόν, ίσες ευκαιρίες, εκτίμηση είναι οι βασικές αρχές για την αναπτυξιακή συνεργασία τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες για την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν στην επιστολή σας η επόμενη πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε να υπογράψετε εταιρικέ σχέσει χρησιμοποιώντα όλα τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σα. Για τον λόγο αυτό, λέει στην επιστολή τη, θα πρέπει να προσαρμόσετε την ανεπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου στόχου Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση τη μετανάστευση. Και εδώ μπαίνουμε σε πολύ ευαίσθητα χωράφια. Πώ ερμηνεύετε εσεί αυτή τη φράση και πώς θα αποφύγουμε να έχουμε μια πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα πιέζει τους εταίρους μας πριν λάβουν απτυξιακή βοήθεια να δεχτούν όλες τις δικές μας ερεσιμότητες για το θέμα της μετανάστευσης. Τι έχετε σκοπό να κάνετε εκεί. Όπως ήδη απάντησα γιατί πιστεύω πως αυτή ήταν και η πρώτη ερώτηση που έλαβα. Θεωρώ πως υπάρχει μια σχέση μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και πολιτικής και μετανάστευσης. Και αυτό έχει να κάνει με τα βασικά αίτια που την προκαλούν. Ξέρετε πως σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα οι σειράξεις, ε, οδηγούν ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Χρειάζεται να φύγουν αλλού. Γιατί, γιατί να γιατί θέλουν να μείνουν ζωντανοί. Η προσωπική μου άποψη λοιπόν είναι πως πρέπει να συνεχίσουμε ε, με την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες, τις χώρες προέλευσης, αλλά και με τις υπόλοιπες. Γιατί γνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στην Ευρώπη, άρα λοιπόν δεν συνεργαζόμαστε μόνο με εκείνες τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, <laughs> So I want to be honest. Um, I think it's not possible. Αλλά επειδή είμαι τίμιο άνθρωπο, να σας πω πως δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους αιρεσιμότητε οι οποίε θα μα επιτρέψουν να πάυσει η μετανάστευση. Αυτό είναι αδύνατον. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε τις ε, οικονομικές ροέ προς τις ε, χώρες, θα διαπιστώσουμε πως η βοήθεια και η συνεργασία η αναπτυξική είναι μόνο ένα κομμάτι ε, αυτής της ε, οικονομικής ροής. Οπότε θα πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει μία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μία μετασυνεργαστική πολιτική και η αναπτυξιακή συνεργασία θα είναι σκέλος αυτής της πολιτικής. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να αποτελέσουμε το μοναδικό εργαλείο μέσα σε αυτό το πακέτο. Ε, δεύτερη ερώτηση, επερώτηση. Λοιπόν, καταλάβατε καλά αυτό που είπα. Θέλουμε εταιρική σχέση και όχι ε, εκ των άνω εντολές. Γιατί το σενάριο στο οποίο σας αναφερθήκατε δείχνει πως χρειαζόμαστε να κινητοποιήσουμε περισσότερα εργαλεία και εδώ και δεκαετίες ζητάμε το 0,7% του προϋπολογισμού σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των χωρών μας. Και αυτή τη στιγμή μόνο τέσσερις ε, χώρες κράτη-μέλη έχουν φτάσει στο 0,7% σε επίπεδο αναπτυξιακή βοήθειας. Εσείς ήσασταν υπουργό Οικονομικών. Πού είναι το πρόβλημα? Γιατί βλέπουμε τα δημοσιονομικά θέματα ε, μέσα από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βλέπουμε το τι ε, οδηγίες απευθύνουμε στα κράτη τα οποία δεν συμμορφώνονται και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ενδεχομένως ε, και το γεγονός πως δεν επιτυγχάνουν αυτά τα ποσοστά τα οποία έχουμε θεσπίσει. Απάντηση. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. γιατί έχει να κάνει με αποφάσεις που λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο, όχι μόνο στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ξέρω ως πρώην υπουργό Οικονομικός πως το προϋπολογισμό τον καταθέτει στο Κοινοβούλιο το Υπουργείο Οικονομικών. Και από αυτή την εμπειρία που έχω και από εκείνη την οπτική γωνία θα έλεγα πως προσωπικά πιστεύω πως θα έπρεπε οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων θα πρέπει να συζητήσουν αυτό το θέμα του ποσοστού του 0,7% του ΑΕΠ ως αναπτυξιακή βοήθεια. Και εγώ έχω κάθε διάθεση να το κάνω, μπορώ όμως να κάνω μόνο αυτό που μου αντιστοιχεί ίσως μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, γιατί είναι αν είναι αυτή η συζήτηση, μια συζήτηση που περιορίζεται στους υπουργού που είναι υπεύθυνοι για αναπτυξιακή βοήθεια και συνεργασία, τότε κατά τη γνώμη μου δεν φτάνει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στο μέλλον για να δούμε πώς μπορούμε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί οικονομικών να εμπλακούν στη συζήτηση αυτή και έτσι να πιέσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, Μισελ Ριβασί, επόμενη ομιλήτρια, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Οι ερωτήσεις που έχω να κάνω έχουν να κάνουν με τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Γιατί ωραίο είναι να λέμε πως ναι, θα πετύχουμε ε, τους στόχους αν βιώσιμης ανάπτυξη για την Ατζέντα 2030, αλλά αν δεν ε, αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιβάλλοντος δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και βέβαια είναι πάρα πολύ κερδοφόρα αυτά τα διασυνοριακά εγκλήματα. Μετά λοιπόν ε, το λαθρεμπόριο, την σωματεμπορία και τα ανακροτικά είναι το τέταρτο πιο κερδοφόρο ε, διασυνοριακό εμπόριο. Οπότε τι θα κάνετε για να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά στις χώρες τις αναπτυσσόμενες και κυρίως ε, στην λαθροθυρία, ε, ε, στην λαθροαλία ε, και σε όλα τα σχετικά. Είσαστε έτοιμοι να διευρύνετε τις αρμοδιότητες στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας και της αναπτυξής συνεργασίας για να καλύψετε και τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ απάντηση. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Θεωρώ πως Όλοι κατανοούμε τη σημασία που έχει ένα καθαρό περιβάλλον. Τώρα, το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή ή κάποια άλλα στοιχεία που άπτονται αυτής, νομίζω πως το καλύτερο είναι αυτό το καινούριο σύμφωνο που παρουσιάζει η νέα Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σε επίπεδο δημόσιων συζητήσεων που γίνονται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, ε, έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας πολύ ε, στις εσωτερικές διαστάσεις αυτής, αυτού του πράσινου συμφώνου. Αλλά αυτό το Green Deal θα πρέπει να έχει και μια εξωτερική διάσταση. Και αυτό είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και τα θέματα του περιβάλλοντος μέσω της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους. Ξέρω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί πάνω από 20% από τα αναπτυξιακά του κονδύλια, για θέματα περιβαλλοντικά. Αλλά συμφωνώ μαζί σας, χρειάζονται περισσότερο, δεν φτάνει. Για παράδειγμα, μετάβαση στην ε, ε, κυκλική οικονομία και στην μείωση των εκπομπών ρηπογόνων ουσιών και στις χώρες εταίρους. Και τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε εσείς, λαθροϊλοτομία κτλ. Αυτό το Green Deal θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να θέσουμε ε, και στην αναπτυξιακή μας συνεργασία τα θέματα του περιβάλλοντος και μάλιστα να τους δώσουμε προτεραιότητες στις συζητήσεις που έχουμε με τις χώρες εταίρους. Έχουμε ε, ε, επερώτηση. Ναι, αυτό το Green Deal είναι μια πολύ όμορφη φράση, αλλά χρειάζονται κυρώσεις, έλεγχοι. Και θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν κοίταζα την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα τα διατροφικά, είπαμε η χρήση της στις χώρες της αναπτυσσόμενας έχει να κάνει με παραπάνω από 200.000 θανάτους λόγω οξίας δηλητηρίας κάθε χρόνο. Τι θα κάνετε λοιπόν εσείς ως υποψήφια επίτροπος να γνωρίζουμε πως απαγορεύονται αυτά τα εντομοκτώνα στην Ευρώπη για παράδειγμα γιατί είναι πάρα πολύ δηλητηριώδη, είναι τοξικά, αλλά τα εξάγουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν δεν έχουν το οπλοστάσιο για να τα ελέγξουν, για να τα περιορίσουν κτλ. Τι θα κάνετε. Γιατί εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που μας επιτρέπει να μην δηλητηριάζουμε τους ανθρώπους που ζουν στις χώρες αυτές όπου δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να τους προστατεύσουν. Απάντηση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει να έχουμε κυρώσεις και κανονισμούς. Και αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, για τη Γεωργία θα έλεγα πως είναι κομβική, ξέρετε πόσα εκατομμύρια ε, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες ε, παίρνουν το εισόδημά τους από την γεωργία. Αλλά είναι και ένας από τους χώρους που επηρεάζεται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και επίσης είναι και μεγάλος, ε, μεγάλη πηγή ρήπων ε, αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε χρειάζεται μία μετάλλαξη των ε, παγκοσμίων συστημάτων έτσι ώστε τα τρόφιμα που φτάνουν σε 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050 να είναι αυλαβή. Η διατροφική ασφάλεια είναι σημαντική για όλους και για τους Ευρωπαίους και για όλους. Μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε τις αφρικανικές εταιρείες και τις αφρικανικές αρχές, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές ε, ρυθμίσεις, τους κανόνες. Και για παράδειγμα, εγώ με ερευνητικά ε, ιδρύματα ή με άλλους εμπλεκόμενους θα έχω κάθε διάθεση να ε, συνεργαστώ έτσι ώστε να το πετύχουμε αυτό. Λόγω τώρα έχει ο από Είμαι πεπισμένος ότι έχετε προετοιμαστεί πολύ καλά για τα της που θα αναλάβετε και θα ήθελα λοιπόν γι' αυτό μια συγκεκριμένη απάντηση, συγκεκριμένη ερώτηση. Εδώ και κάποια χρόνια ακούμε τη δικαιολογία ότι η αναπτυξή βοήθεια για τους Παλαιστινίους οι οποίοι πολλές φορές έχουν λάβει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικούς σκοπούς και ενέργειες. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι είναι η υπόθεση από το 2012 για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων από συγκεκριμένους ανθρώπους για τρομοκρατικούς σκοπούς. Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έκτοτε, πώς έχει διερευνήσει την περίπτωση και εσείς στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας πώς θα κοιτάξετε αυτήν την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και πώς θα εμποδίσετε τέτοια προβλήματα να ανακύψουν και στο μέλλον. Εάν μπορείτε να μας μιλήσετε για συγκεκριμένα μέτρα ώστε να καταπολεμήσετε αυτό το πρόβλημα και να το εξαλείψετε. Uh, Κύριε Επίτροπε. Ελπίζω και πιστεύω στην διαφάνεια. Πάντοτε, όταν χρησιμοποιούμε το χρήμα, τα χρήματα των φορολογουμένων, θα πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί και ιδιαίτερα διαφανείς. Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε τι πετύχαμε. Γιατί χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων και τι επιτυγχάνουμε με τη χρήση τους. Αυτό είναι και θέμα νομιμοποίησης της δράσης μας. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, στους πολίτες, τι επιτυγχάνουμε, ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των προγραμμάτων μας αναπτυξιακής ε, συνεργασίας και ανάπτυξης. Από αυτήν την προοπτική λοιπόν είμαι ε, πλήρως ταγμένη στο σκοπό της, ε, στο στόχο της διαφάνειας και είμαι αποφασισμένη να κάνω περισσότερα και όσο μπορώ καλύτερα στην, ε, ε, στο μέλλον. Το συγκεκριμένο σχέδιο που αναφέρατε στην ερώτησή σας πρέπει να το διαβάσω καλύτερα. Δεν γνωρίζω πολύ καλά τα στοιχεία. Διάβασα πολύ εντατικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν τα ξέρω όμως όλα ακόμα. Αλλά θα φροντίσω να επανέλθω με μια συγκεκριμένη απάντηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επερώτηση. Ευχαριστώ. Πολύ καλό που λέτε ότι μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά ήθελα λίγο να εμβαθύνουμε στην προηγούμενη ερώτησή μου. Και να θέσω μια επιπλέον ερώτηση. Προφανώς υπάρχουν δις από αναπτυξιακή βοήθεια που πηγαίνουν προς την Παλαιστινική Αρχή αλλά δεν έχουν πάντοτε θετικές συνέπειες. Δεν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει εδώ κατάχρηση και να υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία να το ε, ε, διερευνήσουμε. Μήπως χρειάζεται ένα εναλλακτικό μοντέλο αναπτυξιακής βοήθειας σε αυτή την περιοχή για να πάυσει αυτή η κατάχρηση των ε, διεθνών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αλλού από την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτή η σύραξη κρατάει δεκαετίες. Θα πρέπει λοιπόν να πάψει αυτή η ένταση, η συνεχιζόμενη ένταση και η διάθεση των ανθρώπων να φύγουν από την ε, χώρα τους. Τι θα κάνετε εσείς στη διάρκεια της θητείας σας για το θέμα αυτό. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Νομίζω όλοι επιθυμούμε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτός ο απότερος στόχος μας. Μια πτυχή που με απασχολεί είναι πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερες γυναίκες και τους νέους στην ειρηνευτική διαδικασία. Όπως είπα νωρίτερα, έχω εργαστεί ως ειδική αντεταλμένη για θέματα διαμεσολάβησης για την ειρήνευση. Σε αυτό το ρόλο μου αναζητούσα πρωτοβουλίες για το πώς να προσελκύσουμε τους νέους και τις γυναίκες στις προσπάθειες για ειρήνευση. Διότι αν τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναλάβουν κάποιο ρόλο, αυτό μπορεί να διευκολύνει και την επίτευξη των στόχων. Να και ένα ακόμα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε τη δημιουργία ειρήνης στο ασταθές περιβάλλον μας. Μάλιστα. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπεάτα Κέμπα από το ECR. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία υποψήφια, για αυτά που είπατε, που μας δημιουργούν ελπίδα για νέα και νέα ποιότητα στη συνεργασία. Είπατε εταιρική σχέση και όχι επιταγές, όχι εντολές άνωθεν. Είναι πολύ σημαντικό για τη διεθνή συνεργασία ιδιαίτερα για τις χώρες που η κατάσταση είναι πολύ κακή και πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και τη συνεργασία. Έχω μια ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας. Το θέμα είναι, είναι αποτελεσματικές οι δράσεις μας, ιδιαίτερα στις χώρες προέλευσης, από τις χώρες προέλευσης μεταναστών. Γιατί ε, είχαμε πολλές αποστολές σε πολύ δύσκολες ε, στιγμές, ε, ιδιαίτερα για το θέμα της διαχείρισης μετανάστευσης. Μεγάλο τμήμα της αναπτυξιακής συνεργασίας ε, γίνεται έμεσα. Ε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει σε άλλους φορείς ε, την παροχή της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ή φορείς εκτέλεσης ε, αναλαμβάνουν την εκτέλεση αυτής της βοήθειας. Οπότε, ερωτώ το εξή. Θα χρησιμοποιήσετε και την εμπειρία πιο μικρών χωρών μελών και όχι μόνο των μεγαλύτερων χωρών μελών, γιατί στα πλαίσια τη κοινωνία των πολιτών οι μη κυβερνητικέ οργανώσει δεν έχουν την ευκαιρία συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Όμω έχουν μεγάλες, ε, μεγάλη και πλούσια εμπειρία σε ό,τι αφορά την ε, μετανάστευση. Έχετε σκοπό να αφογκραστείτε και τις χώρες αυτές, τις μικρότερες. Η Επίτροπος, η υποψήφια Επίτροπος. Σαφώς ε, και είμαι πρόθυμη να μάθω περισσότερα, είμαι πανέτοιμη και πρόθυμη να συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη. Φυσικά αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και είπα και προηγουμένως ότι δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα να κάνουν το έργο τους. Θα πρέπει να εμπλέξουμε ενεργά και τα κράτη-μέλη και να κάνουν κτήμα τους αυτή την προσέγγιση και τη διαδικασία. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και εταιρικέ σχέσεις. Και γι' αυτό ο διάλογος και οι εταιρικέ σχέσεις ε, θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα αν λάβω την έγκρισή σας. Από την προσωπική μου εμπειρία γνωρίζω ότι η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επιτελούν εξαιρετικό έργο σε, σε πολύ εύθραυστες καταστάσεις σε περιοχές και χώρες και είμαι διατεθειμένη να συνεργαστώ και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και με άλλους ενεχομένους και φυσικά να διδαχθώ από την πείρα τους από όποια χώρα και αν προέρχονται μεγαλύτερη ή μικρότερη. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν προτίθεστε να υποβάλλετε έκθεση ε, ανοιχτή δημόσια έκθεση για την αποτελεσματικότητα των δράσεων και την αποτελεσματικότητα ε, της χορήγησης των κονδυλίων. Θα πρέπει να συνδέσουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων της αναπτυξιακής βοήθειας με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης μετανάστευσης. Φτάνουν όντως τα κονδύλια στα μέρη για τα οποία προορίζονται και κυρίως για τις χώρες που είναι πηγές προέλευσης μεταναστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Σίγουρα η παρακολούθηση και η συνεχής επίβλεψη της κατάστασης είναι πολύ σημαντική. Σε ό,τι αφορά τις πιο τροτές περιοχές, Ήδη συναντήθηκα με τον αρμόδιο συνάδελφο για τη διαχείριση των κρίσεων και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά, γιατί διαπιστώνουμε ότι το πρόγραμμα Nexus που αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο να λειτουργεί, έχει αποφέρει καρπούς και θετικά αποτελέσματα. Αλλά φυσικά έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας. Και αυτός είναι ένας τομέας μόνο όπου η συνεργασία θα αποφέρει καρπούς και επιτεύγματα. Και έχετε και προσωπική πείρα στον τομέα αυτό και πολύ ευχαρίστως αν μου επιτρέπετε θα αξιοποιήσω και τη δική σας εμπειρία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Μιγγέλ Ουρμπαν Κρέσπο από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, με ενδιαφέρει και θα συνεχίσω την ερώτηση για την ε, αλληλεπίδραση ανάπτυξης και μετανάστευσης, από διαφορετική σκοπιά όμως. Νομίζω ότι το μείζον σφάλμα και το ναυάγιο της προηγούμενης επιτροπής ήταν η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, της κακώς αποκαλούμενης ε, προσφυγικής κρίσης, αλλά ήταν ε, κρίση δικαίου περισσότερο, γιατί η αναπτυξιακή πολιτική ήταν σημαντική για τη δημιουργία μιας ε, Ευρώπης φρούριο, που είχε εξωτερική διαχείριση των συνόρων και έθεσε την αναπτυξιακή βοήθεια ως όρο προϋπόθεση και ε, προαπαιτούμενο ε, της διαχείρισης της μετανάστευσης ή μάλλον την, την μετανάστευση ως προαπαιτούμενο της χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας. Το θέμα, η υπόθεση της Νιγηρίας είναι του Νίγηρα είναι σημαντική. Θα εξαρτηθεί επίσης η, η, θα, εξαρτη, θα συζητηθούν αντίκτυπος, θα συζητηθεί ο αντίκτυπος αυτής της πολιτικής στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών. Ό,τι και αν κάνουμε και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τηρεί το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου. Και είμαι υπέρμαχος αυτής της προσέγγισης. Και αυτό θα κάνω και ως ε, επίτροπος, αν με εγκρίνεται. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν πιστεύω ότι μόνο η αιρεσιμότητα θα λύσει τη μεταναστευτική κρίση ή γενικώ τη μετανάστευση. Αν ε, πάρουμε το παράδειγμα του Νίγηρα ή άλλων αφρικανικών χωρών, εκεί η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα μικρό κλάσμα των χρηματοπιστωτικών ροών προς τη χώρα αυτή. Και δεν νομίζω ότι αν ε, κλείσουμε τη στρόφιγγα της αναπτυξιακής βοήθειας ε, θα καταφέρουμε να ασκήσουμε επιρροή στην κατάσταση της χώρας. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα η αναπτυξιακή βοήθεια των οικονομικών γενικώ. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είναι ενιαία η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει μια ενιαία πολιτική και η αναπτυξιακή συνεργασία και η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα, ένα τμήμα του πακέτου αυτού του μεταναστευτικού. Αλλά ένα μόνο τμήμα, όχι το σύνολο. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι σαφές. Επερώτηση. Μία κοινότητα αξιών που μετατρέπει τη Μεσόγειο σε ένα υγρό τάφο ή το Σαχέλ σε μεγάλο τάφο, τι κοινότητα αξιών. ο Νίγηρας ε, λαμβάνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο αναπτυξιακή βοήθεια και είναι η φτωχότερη χώρα της Αφρικής. Οπότε έχουμε αποτύχει στην, ε, στον έλεγχο της αναπτυξιακής βοήθειας στη διαχείρισή τη. Τώρα, ο νέο μηχανισμό ε, γειτονία ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία που εξετάζεται, συζητάται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, στόχο έχει ουσιαστικά το μεταναστευτικό έλεγχο, ερωτώ. Γιατί το να θέσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια ως όρο της προηγούμενης διαχείρισης μετανάστευσης είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χωρών προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Ερωτώ λοιπόν, θα τη διακόψετε αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια. υποψήφια Επίτροπος. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πάντα να σώζει ζωές. Αυτή είναι η αποστολή μας, το καθήκον μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την αναπτυξιακή συνεργασία. Γιατί γνωρίζουμε ότι πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι διαβίουν σε συνθήκε εξαθλίωση. Και γι' αυτό έχουμε την αναπτυξιακή συνεργασία για τον κόσμο, όχι για τι κυβερνήσει, για τις κοινωνίε, για τον ιδιωτικό τομέα. Για τον κόσμο, για του πολίτε, για το λαό. Αυτή είναι η δική μου δέσμευση. Και θα κάνω ό,τι μπορώ θα βάλω τα δυνατά μου για να αυξήσω τους οικονομικούς πόρους των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Και έχουμε δεσμευθεί στο 0,15-0,2 μέχρι στιγμής τη επίσημη αναπτυξική βοήθειας, αλλά ακόμη δεν το έχουμε πετύχει ούτε καν αυτό. Και αυτό θα πρέπει στο μέλλον να το αναβαθμίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων με 18 ερωτήσεις. Το λόγο έχει η κυρία Γιουρκεβιτσένε από το ΕΛΚ. Βρήκα πολύ θετική την πρόθεσή σας να συνεργαστείτε με εμά με το Ευρωκοινοβούλιο, στενά. Γι' αυτό ήθελα να μου πείτε, αγαπητή Γιούτα, για την ε, πολιτική σας δράση. Η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει τη μετάβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από δύσκολου καιρού και δύσκολε καταστάσει σε μια νέα κατάσταση. Και στο εξωτερικό, εσείς αναλαμβάνετε τη μεταναστευτική πολιτική, την ενεργειακή συνεργασία με τι κοινωνίε των πολιτών ε, στον υπόλοιπο πλανήτη και την πολιτική γειτονία στη σχέση μα με τη Ρωσία. Τι ε, ρόλο θα, τι δράση θα αναλάβετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι αναπτυξιακή μας συνεργασία και τα εργαλεία ε, της διεθνούς Βοήθεια, θα μα επιτρέψουν να διαφυλάξουμε τι θεμελιώδει αξίες τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου, τη καλή διακυβέρνηση καθώ και της ε, πυρηνικής ε, ασφάλεια, καθώς και τα πρότυπά της, στην ευρωπαϊκή γειτονία και διεθνώ Θα κοιτάξετε το Ευρωκοινοβούλιο να συμβάλλει στη διατήρηση τη ειρήνης και σε περίπτωση που υπάρξουν παραβιάσεις όλων αυτών των θεμελιωδών αρχών, θα κοιτάξετε να υπάρξει και αναστολή της παροχής βοήθειας. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση και σαφώς μπορείτε να με αποκαλείτε Γιούτα. Καμία αντίρρηση. Όπως είπα νωρίτερα σε αυτή την ακρόαση, πρέπει να σεβόμαστε τις εξή αξίες. Θεμελιώδη δικαιώματα, κράτο δικαίου, σε ό,τι και αν κάνουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Για μένα, ως υποψήφια επιτροπεύω για τις διεθνείς μας σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία, σημαντικό θα είναι να βελτιώσω τον σεβασμό κράτους δικαίου και, του κράτους δικαίου και των θεμελιδών δικαιωμάτων μέσω της αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μηχανισμό Γειτονία Ανάπτυξη και Διεθνού Συνεργασία, ενδίκη Έχει πολύ νόημα να έχουμε αυτό το καινούργιο εργαλείο, διότι προ στιγμή έχουμε πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά μαζί με το NDK μπορούμε να τα συγκεφαλαιώσουμε όλα. Και θα είναι μέρος του προπολογισμού μέσω τη νέα μα διοργάνωση. οπότε έτσι θα έχει και περισσότερη εξουσιοδότηση να λάβει θέση εδώ το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα είναι θετικό αυτό ότι θα μπορεί και το Κοινοβούλιο να επηρεάσει τα πράγματα. Πάντω, προσωπικός και από την δική μου προσωπική εμπειρία ω Υπουργό Οικονομικών, με ένα εργαλείο με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μπορούμε να είμαστε συνεκτικότεροι, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι και βεβαίω. Θα είναι μάλλον και απλούστερο να κατανοήσουμε τη δουλειά μας από την σκοπιά των ε, συνεργατών μας. Είμαι λοιπόν πλήρως ε, πρόθυμη ε, και με ενδιαφέρει να δούμε αυτό το εργαλείο στη δουλειά μας. Επερώτηση. Όπως τα γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο πρόκειται να ξεκινήσει διαθεσμικές διαπραγματεύσεις, για το ΕΝΤΙΚ. Ωστόσο, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει μόνο μέρο τη διαπραγματευτική εντολή. Υπάρχει περίπτωση η χθεσινοβραδινή απόφαση του Συμβουλίου για δύο σοβαρέ πτυχέ του εργαλείου αυτού για το Ευρωπαϊκό Αναπταξιακό Ταμείο και τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Γειτονίας Υπάρχει περίπτωση να το επηρεάσει αυτό και οι μελλοντικέ σχέσει να διαμορφωθούν διαφορετικά εάν το Συμβουλίο δεν συμπεριλάβει αυτά τα δύο σκέλη στον κανονισμό του Εντίκη. Πώ θα διαρθρωθούν τα σημερινά αναπτυξιακά εργαλεία ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι, Κοινοβούλιο, ε, Συμβούλιο και οι εταίροι μα. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, όπως είπα νωρίτερα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι καλό είναι να συναρμόσουμε διαφορετικά ε, αναπτυξιακά εργαλεία μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο νομίζω ότι είναι συνετό να ενταχθεί στον ε, τακτικό προπολογισμό για να έχετε κι εσείς περισσότερο λέγει να δω περισσότερη εξουσία οι ευρωβουλευτές. Πάντως, είμαι αρκετά έμπειρη στην πολιτική ώστε να μην μ' αρέσουν οι προβλέψεις και οι υποθέσεις. Δεν θέλω να προδικάζω ότι μπορεί να συμβεί εάν. Εάν βεβαίως ε, εγκριθώ ως Επίτροπος, ε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να καταλήξουμε σε μια κοινή ε, αντίληψη με όλα τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει όμω να δούμε και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι σε κάθε περίπτωση το NDK θα είναι ένα κομμάτι του ευρύτερου αυτού συνόλου. Και τώρα ο λόγος στο Μάρκ Ταραμπελά από τους σοσιαλιστές. Κυρία υποψήφια επίτροπε, κυρία Ούρπι Λάινεν, για την συνοχή των επτεξιακών πολιτικών πρέπει να πούμε ότι οδηγούμαστε στην εξή αξιωματική απέτηση. Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει κάποιο αποτέλεσμα στις χώρες ε, τις αναπτυσσόμενες. Και στο άρθρο 208 αναφέρεται στη συνθήκη ότι πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να κοιτάξουμε να περιορίσουμε τη φτωχιά, των, την, τις αρρώστιες και αυτό θα πρέπει να αποτελεί στόχο των εμπορικών, κοινωνικών, αγροτικών μας πολιτικών ε, και ούτω καθεξής. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης λοιπόν είναι βασική προϋπόθεση η επιδίωξή τους όμως δεν γίνεται βάσον, βάση ε, μηχανισμών αξιολόγηση που είναι αρκετά αξιόπιστη. Στα πλαίσια του ρόλου σα ω Επιτρόπου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τέτοιο είδους πρόθεση τη ανάπτυξη σε όλα τα σκέλη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πώς βλέπετε την συνοχή αυτού του σκέλους της ανάπτυξης στις πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα τον εσείς στο ρόλο σας ως Επιτρόπου, ε, πώ θα επηρεάσετε τα εμπορικά θέματα και αν θα φροντίσετε να υπάρξουν μηχανισμοί που να επιτρέπουν να ελέγξουμε την συνεκτική επιδίωξη των στόχων της αναπτυξιακή βοήθεια. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, ευχαριστώ. Τη βρίσκω κέρια την ερώτηση και βεβαίω έχει να κάνει και με τους στόχους της χελιετία, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την ατζέντα του 2030. Όπως είπα σήμερα ήδη, Για μένα η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια πηξίδα, ένας μπούσουλας. Και θα πρέπει να είναι το πλαίσιο για όλη μας την αναπτυξιακή βοήθεια. Όμως σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχετε και δίκιο. Διότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η, αριστερά, η δεξιά να γνωρίζει τι πει η αριστερά της. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα δούμε τα πράγματα μεμονωμένα. Αν θέλουμε να επιτύχουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη στι γειτονικέ μα χώρε, πρέπει και το εμπόριο να επιδιώξουμε, να προωθήσουμε και τη γεωργία. Όλα αυτά πρέπει να είναι μέρο τη ίδια προσέγγιση. Βεβαίω, η συνεργασία με τον Επίτροπο επί των Εμπορικών, επί Γεωργίας, είναι συνάδελφοι με τους οποίους θα πρέπει να συζητάμε για να υπάρχει συνοχή στο έργο της Επιτροπής. Ένα εργαλείο προς αυτό το σκοπό θα ήταν ίσως οι εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές που προσπαθούμε να επιμείνουμε ότι οι εταίροι μας θα πρέπει να τις σχεδιάσουν και θα πρέπει και να τους στηρίξουμε για να έχουμε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση και να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Επερώτηση. Οι πρόσφατε αξιολογήσει έδειξαν ότι οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τι αναπτυσσόμενε χώρε δεν παίζουν αρκετά ε, καλό ρόλο στην αξιολόγηση και την ε, υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Πώ θα συνεργαστείτε με του απεσταλμένου μα ώστε να βεβαιωθείτε ότι η επιδίωξη των στόχων μα είναι στην πρώτη γραμμή τη δουλειά και τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Είδα επανειλημμένο τον κύριο Μπορέλ, είπα το εκπρόσωπο και, και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι χαρά μου που θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Βλέπω ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να ενταχθεί και στις εξωτερικές μας σχέσεις και υποθέσεις. Άποψή μου λοιπόν είναι ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα πρέπει να κάνουμε μια κοινή ερμηνεία των πραγμάτων, του διεθνούς προσκυνήου και του τι συμβαίνει στον κόσμο, μετά να καταρτήσουμε μια κοινή στρατηγική που να βασιστεί σε αυτή την ερμηνεία, σε αυτή τη μελέτη και μετά να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, να τα εντάξουμε και να τα προωθήσουμε, να τα διοχετεύσουμε στις λεπτομέρειες των προγραμμάτων μας. Είμαι λοιπόν ε, πρόθυμη να συνεργαστώ με τον πατό εκπρόσωπο και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Από τη Ρηνιού η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. Καλημέρα σας. Εδώ είμαι, κυρία Ορπιλάιν. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε γυναίκα ε, υποψήφιο για το θέμα της, ε, του χαρτοφυλακίου ανάπτυξης. Βλέπω από τις απαντήσεις σας πως ε, η ισότητα μεταξύ ανθρώπων είναι προτεραιότητα για σας με προτεραιότητα επίσης τη μάχη κατά της βίας κατά των γυναικών, όπως επίσης και υπέρ της ισότητας στην εκπαίδευση για τη γυναίκα. Επίσης, τι γίνεται με την πρόσβαση ε, στην ε, αντισύλληψη, στην αναπαραγωγική υγεία και τι θα γίνει επίσης με κάποια άλλα ε, θέματα που αποτελούν κατάφορη παραβίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά θίγουν επίσης και τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, στο μέλλον και στην υγεία. Εσείς πώς θα θέσετε σε εφαρμογή αυτές τις δεσμεύσεις σας, ποια πολιτικά μέτρα θα λάβετε για να συζητήσετε τα θέματα αυτά με τις χώρες εταίρους και τι θα κάνετε με την κοινωνία των πολιτών η οποία έχει αναλάβει δράση υπέρ αυτών των δικαιωμάτων. Κύριε Ψήφια Επίτροπος, ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ ε, για μια τόσο σημαντική ερώτηση. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι θέματα τα οποία θα είναι κεντρικά στις προσπάθειες που θα κάνουμε για να πετύχουμε την ισότητα των ε, ε, φίλων. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα και μια και έχω την ευκαιρία θα ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μίμητσα για τις προσπάθειες που έχει κάνει για τα θέματα της ισότητας των φύλων να σας πω πως έχουμε ε, την πρωτοβουλία Spotlight που είναι σημαντική και σίγουρα επιθυμώ να συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση και στο μέλλον. Επίσης θεωρώ πως ε, για την ισότητα των φίλων και τις ίσες ευκαιρίες χρειάζεται μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση σε όλο το κόσμο, να συνεργαστούμε με διεθνείς οργανισμούς, με την κοινωνία των πολιτών, με τις εθνικές κυβερνήσεις, γιατί μόνο μέσω της συνεργασίας θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα. Κάτι που είναι σημαντικό για όλους, όχι μόνο τους Ευρωπαίους, αλλά και για τους πολίτες του υπόλοιπου κόσμου, είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. Και εκεί χρειάζεται να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις επιδόσεις μας. Εγώ είμαι γυναίκα επίτροπος και για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση υπηρεσίες υγείας ε, θεωρώ πως είναι θεμελιώδες δικαίωμα για όλους μας και θα έπρεπε το ίδιο να ισχύει και στις ε, ε, χώρες εταίρους μας. Επερώτηση. Στην απάντησή σας αναφερθήκατε επίσης ένα ενδεχόμενο ε, σχέδιο δράσης για τα φύλλα. Αν δεν κάνετε το Gender Plan 3, ε, που θα μπορούσε να είναι αυτό το σχέδιο δράσης. Τι εργαλείο μπορείτε να προτείνετε για να συνεχιστεί η στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και η ισότητα μεταξύ ανθρώπων είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ. I can in the front of the... Θα σας υποσχεθώ εδώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πως το σχέδιο δράσης υπαριθμών 3 για την ισότητα των φύλων θα γίνει πραγματικότητα. Ε, αναλαμβάνω αυτή τη δέσμευση και θα το πραγματοποιήσω. Είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό για μας για να προσφέρουμε ε, και να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ των φύλων. Ε, από το ΕΛΚ ο Λούκας Μαντελή είναι ο επόμενος εισηγητής. Ε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας εγχαρώ για την υποψηφιότητά σας και να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε σήμερα και τη δέσμευση με την οποία αναφερθήκατε ε, στη βασική αρχή. Ο άνθρωπος θα πρέπει να στηρίξει τον άνθρωπο ε, στα δικαιώματα τα ανθρώπινα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια τεχνική ακρόαση, βλέπουμε ποιε είναι οι πολιτικέ σα προτεραιότητε, αλλά βλέπουμε και την ανθρώπινη διάσταση. Καταλαβαίνετε πω όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οικονομία γιατί οι ευκαιρίες που προσφέρουν στους ανθρώπους μας έχουν να κάνουν με την οικονομία. Γιατί όταν υπάρχει η σφριγιλή και στεναρή οικονομία, πολλά μπορούν όλοι να πετύχουν. Έχουμε το, την παιδεία και το κράτος δικαίου, ε, ακόμα και για τα θέματα της τεχνικής παιδείας, γιατί από εκεί προέρχονται όλες οι ευκαιρίες. Τι θα κάνετε λοιπόν για να ενισχύσετε την κατάρτιση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό πρέπει να το προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η υποψήφια επίτροπος, όπως είπα και στην ε, ε, εισαγωγική μου παρουσίαση ήμουν δασκάλα πριν γίνω επίτροπος. Οπότε στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως διδακτικό προσωπικό είδα πώς η εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει ζωές. Και διαπιστώνω πως θα πρέπει να αναλάβουμε τη δέσμευση και εγώ είμαι πρόθυμη να το κάνω, να χρησιμοποιήσουμε μέσω του NDK αυτό το 20% της χρηματοδότησης δηλαδή για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό για μένα. Τώρα, τι με ανησυχεί. Η ποιότητα της παιδείας που θα προσφέρουμε, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόσβαση στην παιδεία, έχει να κάνει και με την ποιότητα της προσφερόμενης παιδείας. Πρόσφατα λάβαμε μία έκθεση της Παγκοσμίου Τράπεζας και το μήνυμα στην έκθεση αυτή είναι πως δυστυχώς πολλοί άνθρωποι παρόλο που συμμετείχαν ε, στην παιδεία ακόμα δεν μπορούν ούτε να μετρήσουν ούτε να διαβάσουν. Οπότε αυτό που θα τόνιζα περισσότερο και θα χρηματοδοτούσα πιο πολύ και το οποίο θα τόνιζα πιο πολύ είναι η ποιότητα της παιδείας που προσφέρουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα προσωπικά είναι ξεκάθαρο πως η παιδεία είναι το κλειδί για να μειώσουμε ε, την φτώχεια. Άρα λοιπόν αποτελεί για μένα μια προτεραιότητα. Ε, Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μπήκατε σε βάθος στα θέματα αυτά. Ίσως είναι και πολιτιστικό το ερώτημα όταν μιλάμε για ισότητα των φίλων, για το κατά πόσο οι... τα κορίτσια έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα γόρια όταν είναι παιδιά ή ακόμα και όταν είναι ενήλικες, όταν μιλάμε για τα θέματα τα εκπαιδευτικά. Άρα λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε σε ποιους κλάδους και με ποιους άλλους επιτρόπους θα συνεργαστείτε έτσι ώστε να ε, ανταποκριθείτε στην υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσουμε και άλλα μέρη στον πλανήτη μας με τις ευρωπαϊκές αξίες που είναι ε, ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες και βεβαίως και στον χώρο της παιδείας και στις ευκαιρίες που θα έχουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε για την ποιότητα. Η ποιότητα χρειάζεται καλούς καθηγητές και αυτό το γνωρίζετε μια και εσείς η ίδια είστε διδακτικό προσωπικό. Η υποψήφια επίτροπος βεβαίως και με την Επίτροπο για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά η προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλη τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή σε όλο το σώμα της Επιτροπής. Πρόσφατα πήγα σε ένα ε, ε, στρατόπεδο προσφύγων στην καμπέλα της Ιθοποιίας. Και με άγγιξε πολύ βαθιά αυτή η εμπειρία γιατί εκεί ε, στεγάζονται πάνω από 50.000 άνθρωποι και κάτι το οποίο βρήκα ιδιαίτερα λυπηρό ήταν πως μόνο το ίμιση των παιδιών εκεί πάνε σχολείο. Από αυτή την άποψη λοιπόν και το έχω συζητήσει με, τους, με, τον Επίτροπο για την διαχείριση κρίσεων, πως θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για την πρόσβαση στην παιδεία των ε, κοριτσιών και των γυναικών και στα στρατόπεδα προσφύγων. Γιατί είναι σημαντικό και οι άνθρωποι αυτοί που ζουν εκεί να έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Πιέρ Φρανσέσκο Ο Πιέρ Φραντσέσκο Μαγιορίνο από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επιψήφια Επίτροπο. Θα συμφωνήσω με πολλά από όσα υπόθηκαν, απλώ θέλω να σταθώ στο εξή πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε τη μετατόπιση της απόδοσης στόχων από την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις ε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον έλεγχο των συνόρων, για, την, ε, για τον έλεγχο των μετακινήσεων στον πλανήτη. Και χωρίς σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε με κοινοβουλευτική λογοδοσία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκε για αυτόν τον σκοπό ήταν των καταπιστευμάτων. Ε, μια πολύ ευέλικτη δομή η οποία όμω υπέκρυπτε, πιστεύω, την αδιαφάνεια, την αμφισημία στη χρήση του. Δηλαδή το 2018 ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκε η Λιβική Ακτοφυλακή, που καμία σχέση δεν έχει με αναπτυξιακή συνεργασία για την ανάπτυξη γενικότερα. Υπό αυτήν την έννοια θέλω να σα ρωτήσω τι άποψη έχετε για τα κονδύλια και το τι γίνεται με τα καταπιστεύματα και το πώ χρησιμοποιούνται. Τι θα πρέπει να αλλάξει εδώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε και τη χώρα διέλευσης μεταναστών ή προσφύγων. Γιατί 85% των μεταναστών προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες ή διαμένουν σε αναπτύσσόμενε χώρες και μέσω της αναπτυξιακή συνεργασίας μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτές τις χώρες και τις χώρες προέλευση, δηλαδή, αλλά και τις χώρες διέλευση μεταναστών. Γνωρίζω ότι το Αφρικανικό Καταπιστευματικό Ταμείο είναι ζήτημα που διχάζει κάπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπα και νωρίτερα πάντως, η διαφάνεια κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική αξία και αντιλαμβάνομαι ότι και στο μέλλον, όταν συζητούμε το μέλλον του καταπιστεύματος για την Αφρική ή γενικώ ε, το μέλλον των καταπιστευματικών ταμείων, στη συζήτηση αυτή θα πρέπει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν γνωρίζω ακριβώς ε, τα σχέδια. Πάντως σίγουρα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον για τα θέματα αυτά. Επερώτηση. Οπότε, μάλλον θέλω να, να εμείνω σε αυτό το σημείο και να αντιληφθώ κατά πόσον συμφωνούμε πρέπει να συμμετέχει ε, το Ευρωκοινοβούλιο σε συμβουλευτικό ρόλο για να εξασφαλίζει τον έλεγχο και το πώς χρησιμοποιούνται ε, τα κονδύλια από τα καταπιστεύματα, ότι λειτουργούν συνεπώς και από την άλλη να βλέπουμε κατά πόσο μπορεί να είναι ασύμβατες κάποιες δράσεις, κάποιες χρηματοδοτήσεις εργαλεία, όπω η χρηματοδότηση τη λιβική εκτοφυλακή. Δεν έχει αυτό σχέση με τα καταπιστεύματα. Δεν υποστηρίζουμε έτσι την χώρα διέλευση, που είναι σημαντικό θέμα και σωστά το θίξατε. Απλώ χρηματοδοτούμε εργαλεία για να μπλοκάρουμε τα σύνορά μα και για να, εξωτερικό, ε, να αναθέσουμε εξωτερικώ την φύλαξή του. Υποψήφια Επίτροπος. Η συνοχή των πολιτικών μας έχει κέρια σημασία. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνοχή των πολιτικών μας. Παντού. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για 16 χρόνια ήμουν μέλος της Φιλανδικής Βουλής και πραγματικά τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για το έργο σας. Εσείς είστε άμεσα εκλεγμένοι από το λαό. Εμένα με διόρισαν, ε, θα με εγκρίνετε εσείς αν το κάνετε. Αλλά εσείς είστε άμεσα αιρετοί, εκπρόσωποι του λαού. Οπότε εκπροσωπείτε απευθεία τους ε, πολίτε σα. Οπότε τρέφω μεγάλο σεβασμό ε, και εκτιμώ ιδιαίτερο στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα δούμε τι πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε για να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Πιερέτ Χαρισμπέργκερ Φοφάνα. Behind you. Bonjour, Madame la... Πίσω σας βρίσκομαι, πίσω σας. Bonjour, Madame la... Καλημέρα σας, κύριε υποψήφια επίτροπε. Ε, η επιστολή αρμοδιοτήτων των καθηκόντων που σας έστειλε η κυρία Προ, ε, εκλεμένη πρόεδρος ε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική σχέση με την Αφρική και σε εμπορικά ζητήματα. Και απότερο στόχο είναι η δημιουργία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο υπήρων η εξαγωγή ε, ε, φθηνών γαλακτοκομικών προϊόντων προς τη Δυτική Αφρική δείχνει το σοβαρό κίνδυνο που θα ενείχε μία απελευθέρωση τη εμπορία χωροτικών προϊόντων που καταστρέφει πολλές φορές την τοπική παραγωγή, την ε, τοπική γαλακτοπαραγωγή για παράδειγμα. Κάτι που πλήττει άμεσα τις γυναίκες που, είναι, που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της τοπικής παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, Πιστεύετε ότι οι αφρικανικές χώρες θα μπορούν να λάβουν μέτρα ή θα δικαιούνται να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την βιώσιμη οικογενειακή γεωργία και να την προστατεύσουν απέναντι στο, κίνδυνο τη μαζική εισαγωγή φθηνών γεωργικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέτοια μέτρα προστασία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ποσοτικού περιορισμού των ευρωπαϊκών προϊόντων, των ευρωπαϊκών εισαγωγών, δίνοντα ε, ε, προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα ή θεσπίζοντας φόρους ή δασμούς για διάφορα γεωρικά προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης. Σας ευχαριστώ. Υποψήφια Επίτροπος έχει το λόγο. Και η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών αποτελεί σημαντικό τμήμα των προτεραιότητων μας. Και όλοι όσοι πήγαμε στην Αφρική γνωρίζουμε ότι η Αφρικανική Γεωργία στηρίζεται στις ε, μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Και σίγουρα η τοπική γεωργία, που είναι γεωργία μικρής κλίμακας οικογενειακού χαρακτήρα, είναι σημαντική για την Αφρική. Είμαι έτοιμη να λάβω τα κατάλληλα μέτρα, οπότε η απάντησή μου είναι καταφατική. Και μία πιθανότητα θα ήταν μία ολιστική, σφαιρική στρατηγική για την Αφρική. Αυτό αναφέρεται και στην επιστολή των καθηκών και αρμοδιοτήτων μου. Και σε αυτή την ε, ολιστική σφαιρική στρατηγική για την Αφρική θα πρέπει να περιλάβουμε και τη γεωργία και το εμπόριο και το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οπότε αυτή η σφαιρική στρατηγική θα μας δώσει νέες ευκαιρίες για να στηρίξουμε και την γεωργία στην Αφρική. Και θα είναι ένα νέο εργαλείο που θα έχουμε στη διάθεσή μας προς χρήση. Επερώτηση. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει και με ποια μέτρα ώστε οι ευρωπαϊκές γεωργικές επενδύσεις που γίνονται στα πλαίσια της σύμπραξης ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν θα ε, παρεμποδίσουν τα δικαιώματα των λαών, ιδιαίτερα για την ε, γεωργία και την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα σε μια ε, περίπτωση που επιχειρήσεις ε, πιέζουν τις κυβερνήσεις να χαλαρώσουν τους κανόνες προς, το όφελος, προς όφελος των επιχειρήσεων. Η υποψήφια Επίτροπος. Όταν αναφερθήκατε στον ιδιωτικό τομέα, πραγματικά θέσετε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων και δεν συζητήσαμε ακόμη εκτενώς για το θέμα αυτό. Γιατί αν όντως θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, θα πρέπει να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι απαραίτητο. Η δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό που έχει ήδη γίνει μέσω αυτής της συμμαχίας, της πρωτοβουλίας ε, για την συμμαχία αυτή με την Αφρική του Πρόεδρου Γιουνκέρ. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ήταν ελπιδοφόρα. Πάντως στο μέλλον θα πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις ε, στην Αφρική με ανάμειξη και του ιδιωτικού τομέα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην υποσαχάριο Αφρική θα χρειαστούν 18 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης το χρόνο για να απασχοληθούν όλοι οι νέοι που μπαίνουν στην αγορά εργασία. 18 εκατομμύρια νέε θέσει εργασία θα πρέπει να δημιουργούνται κάθε χρόνο στην υποσαχάρια Αφρική. Οπότε ακόμη και να αυξήσουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, δεν πρόκειται ε, να τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να αναμίξουμε και τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικά κεφάλαια. Φυσικά χρειάζονται κανόνες ε, και διατάξεις. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και τα μέλη και την ε, υποψήφια επίτροπο ότι έχουμε μέχρι στιγμής ολοκληρώσει το ίμιση των ερωτήσεων. Οπότε τα πάμε μια χαρά νομίζω. Αλλά έχουμε 12 ακόμη ερωτήσεις, οπότε δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Η κυρία Ντομινίκ Μπίλντε από, τους, από την ταυτότητα και δημοκρατία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας κυρία μου. Η στρατηγική σας για την Αφρική υποκρύπτει μια σκοτεινή πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά διαπραγματεύσεις για το στάδιο μετά την Κοτόνου αποδυναμωμένη σε σχέση με το τι συνέβαινε στις αρχές της χιλιετίας. Έχουμε νέους πρωταγωνιστές στην Κίνα, τη Ρωσία και το βάρος της διεθνούς οικονομίας αλλάζει ε, διότι φεύγει το, Ευρω... το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κρίση του ευρώ, το Brexit δείχνουν ότι περνάμε μια πολιτική κρίση. Επιπλέον η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μας κάνει να χάσουμε ένα σημαντικό συνεργάτη στο εμπορικό, στρατιωτικό και ειρηνευτικό προσκήνιο, το 15% του ευρωπαϊκού προπολογισμού που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο 2015 έως 2016 ε, και το 2018 ε, είχε επίση προσφέρει το 0,7%. Είχε συμβάλει στην επίσημη αναπτυξική βοήθεια. Και η Γερμανία βεβαίω έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα Marshall από τον Ιανουάριο του 2017 για την Αφρική. Όμω οι προθέσει του G5 και του Σαχέλ δείχνουν ότι οι οικονομικέ δεσμεύσει δεν γίνονται πραγματικότητα πάντοτε, αλλά μένουν λόγια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Έχετε σκεφτεί όλε τι συνέπειε που θα έχει το Brexit στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική μετά την ε, Συμφωνία τη Κοτονού και πώ θα την αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Θα έλεγα σε ό,τι αφορά το Brexit. Όλα αυτά είναι θέματα εθνική κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, τη κυβέρνηση και του λαού του. Όμω, το Ηνωμένο Βασίλειο σαφώ ήταν σημαντικό δωρητή, ιδίω οι με κυβερνητικέ οργανώσει του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν ε, σοβαρότατο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Οπότε, από αυτήν την οπτική γωνία, ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι ένα πολύτιμο συνεργάτη ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και στο μέλλον. Όμω, όπω γνωρίζουμε, τα ερωτήματα που περιβάλλουν το θέμα Brexit είναι πολλαπλά. Δεν είναι η δική μου δουλειά, πιστεύω, ούτε η σημερινή μου αρμοδιότητα να προδικάσω ή να, να πιθανολογήσω για αποτελέσματα. Πάντω η συνεργασία του με τον Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύτιμη και ελπίζω να την συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Μια τεχνική παρατήρηση από πλευράς διερμηνέων. Όταν ρωτάμε τις ερωτήσεις μας και φοράμε τα ακουστικά ε, στο λαιμό, δεν είναι πολύ απλό το. Δεν ακούτε καλά η ερώτηση. Παρακαλούμε να τα βάζετε πάνω στο εδρανό σα, αν θέλετε. Τη στιγμή που κάνετε την ερώτηση και μετά όλα θα είναι τέλεια. Συνεχίζουμε με την επερώτηση. Όταν ρωτάτε την ερώτηση, είναι πολύ κοντά ε, στο μικρόφωνο, μπορείτε να τα κουμπίσετε στο έδρανο. Επερώτηση. Τα, μπλεξα τελείω. Πελάγωσα. Ερώτηση. Το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά τόσα πολλά για την Αφρική δεν εκτιμάται από όλου και προκαλεί και ερωτήσει. Ο Όμιλο Κριστή που ε, συνδέει από έναν Ευρωπαίο διπλωματή λέει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά ένα δι δολάριο Μάλλον η Κίνα ε, δαπανά ένα δις δολάρια και έχει ε, φοβερά αποτελέσματα στην προβολή της, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 20 και καθόλου αποτελέσματα από, σε, σχέση με, σε σύγκριση με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που έχουμε πετύχει, που θέλουμε να πετύχουμε, η προβολή όλων αυτών στην κοινή γνώμη, είναι ένας στόχος εφικτός. Ευχαριστούμε κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Προσωπικός δεν βλέπω να έχουμε χάσει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Το 2018 ως Ευρωπαϊκή Ένωση 14 δις ευρώ δώσαμε στην και βοήθεια και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη ξεπεράσαμε τα 70 τεράστια ποσά και δυστυχώς χρειάζονται κι άλλα. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Γι' αυτό και ανέφερα το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Κατανοώ ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην Αφρική, αλλά θα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να είναι μέρος όλης αυτής της πολιτικής και προσέγγισης. Σε ό,τι αφορά την Αφρική, το μέλλον της Αφρικής είναι και το μέλλον της Ευρώπης. Είναι αλληλένδετες οι δύο ήπειροί μας όμως θέλω να αλλάξει λιγάκι αυτό που ακούγεται συστηματικά στην Αφρική. Έχουμε 1,2 δις ανθρώπους στην Αφρική και η μισή μόνο είναι κάτω των 35, άνω των 35. είναι μια χώρα με ευκαιρίες, μια περιοχή με ευκαιρίες και έχει πολλά θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει και να υποστηρίξουμε. Τα λόγο έχει τώρα ο κύριος ε, Ρίσαρτ Τσαρνέτσκι από το ECR. Κυρία αντιπρόεδρε της κυβέρνησης. Κύριε Υποψήφια Επιτροπέ. Ήθελα να σας πω τα εξής. Γιατί Κάποια θέματα που θέλω να συζητήσουμε εκ μέρου πολιτισμού ομάδα είναι σημαντικά και θα ξεκινήσω λέγοντα κοίτο στα φιλανδικά και μετά θα μιλήσω πολωνέζικα για να έχουμε πολλέ γλώσσε στο κοινοβούλιο. Για πολλά χρόνια ήμουν μέλο τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ. Τώρα μιλούμε για Συμφωνία Οικονομικής εταιρική Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των χωρών ε, και οι συζητήσει ε, είναι σε αρκετά προηγμένο στάδιο. Βέβαια, πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του γιατί αυτή η διαπραγματευτική διαδικασία έχει επιβραδυνθεί και έχει προσκρούσει σε ένα σκεπτικισμό από πλευράς των εταίρων μας, των χωρών ΑΚΕ δηλαδή. Ε, σκοπεύετε να δώσετε ένα νέο δυναμισμό στην ε, διαδικασία αυτή και να επιταχύνετε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Υποψήφια Επίτροπος. Νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι να πετύχουμε μια συμφωνία ε, με τις χώρες ΑΚΕ μετά από αυτή που έχουμε ως Συμφωνία του Κοτονού. Και είπα προηγουμένως πως για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής, της ε, Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, πως τις θεωρούμε πολύ σημαντικού μας εταίρους. Οπότε αν διοριστώ επίτροπος και ξεκινήσω 1η Νοεμβρίου, όπως ελπίζουμε, το θέμα αυτό θα αποτελέσει και την προτεραιότητα στη δουλειά μου, δηλαδή να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις για την μετά το Κοτονού Συμφωνία, βεβαίως με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επερώτηση. Κοίτο. Ευχαριστώ. Then we continue with uh, the next. Uh, Ωραία λοιπόν. Χίλτεγκαρ Μπέντελε από το ΕΛΚ. Ähm, μέρο τη ε, Επιτροπή μα είχε την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να πάει στη Νέα Υόρκη και είδαμε τι μεγάλε προσδοκίε υπάρχουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πώ θέλουμε να προωθήσουμε τι αξίε μα και σε όλε μα τι πολιτικέ. Γι' αυτό ήθελα να μου πείτε σε θέματα αποτελεσματικότητα, κυρίω για τη συνοχή, τη συνεκτικότητα τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Είναι πολλέ οι δράσει των ε, κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια σωστή διοργάνωση τη όλη μα ε, ε, εφαρμογής προγραμμάτων. Πώ μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τις ίδιες ενέργειες με τις ίδιες προτεραιότητες ώστε όλες οι δράσεις κατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιδιώκουν τους ίδιους στόχους ως προς την ανάπτυξη και να είναι και σαφές το τι κάνουμε και να μπορούμε και να το φέρουμε εις πέρας. Κυρία Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, πραγματικά πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική προοπτική διότι χωρίς την ε, συνεκτικότητα, τη συνοχή στην πολιτική, δεν είμαστε σε θέση να επιτύχουμε κανένα από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και όπως είπα νωρίτερα, βλέπω ότι η ατζέντα του 2030 είναι κάποιο είδους πηξίδα. Ένας οδηγός, ένα πλαίσιο εντός το οποίο πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε τα διάφορα επίπεδα δουλειάς μας. Βεβαίως δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν με κοινό προγραμματισμό, κοινό σχεδιασμό, κοινή αξιολόγηση για να μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματά μας. Είναι σημαντικά να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά εργαλεία. Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές στρατηγικές για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μία που έχει η Φινλανδία, γνωρίζω καλά ας πούμε. Καλό θα ήταν να ανταλλάξουμε μεταξύ μας αυτές τις γνώσεις, τα παραδείγματα του τι κάνουν ως τώρα τα κράτη-μέλη. Και να προσπαθήσουμε, αν κάτι καλό υπάρχει, να το κάνουμε κι εμεί. Πάντω έχετε δίκιο. Χωρί τη συνεκτικότητα στην πολιτική και στην Αφρική και στο εμπόριο και στι εξωτερικέ μα σχέσει, δεν μπορούμε να πετύχουμε την, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι το κλειδί. Επερώτηση. Για το NDC λοιπόν, ένα εργαλείο που μας είπατε ότι μπορεί να πάει πολύ γρήγορα και να ε, υλοποιηθεί αμέσως. Όμως μπορεί να μην είναι τόσο σαφές προς τους στόχους και τη στοχοθέτηση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Νομίζω ότι η υποστήριξη του προπολογισμού θα είναι το βασικό εργαλείο του πακέτου και στο μέλλον. Αλλά συμφωνώ όταν χρησιμοποιούμε την υποστήριξη προς τον προπολογισμό, πρέπει να υπάρχει και ένας μεγάλος βαθμός διαφάνειας για να μπορούμε να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη με τα οποία συνεργαζόμαστε. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε είδους κατάχρηση, υπεξαίρεση, οτιδήποτε τέτοιο, πρέπει να ε, κλείσει κλείσει κάνουλα της χρηματοδότησης. Και ξέρω ότι μέσω τη στήριξη του προπολογισμού έχουμε πετύχει και καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι και στο μέλλον θα είναι ένα από τα βασικά μα εργαλεία. Όχι το μόνο, αλλά ένα βασικό εργαλείο στο πακέτο. Η κυρία Ζαμπό από τη Ρινιού. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας πω πως το 2002 ε, είπε ο πρόεδρος Ιράκ και για το πλανήτη μας. Και μετά από τα δραματικά, τα όσα είπαν το περασμένο την περασμένη Τετάρτη, πυρογνώμονε για το κλίμα θα μπορούσαν να πούνε το ίδιο και για τους ωκεανούς μας ε, που τρέφουν ε, τον πληθυσμό μας. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης χάνει οξυγόνο, ε, χάνει ε, θάλασσα, χάνει ε, χώρο, πνίγεται στα πλαστικά, η κατάσταση στη Βαλτική δεν μπορεί να αναστραφεί και είναι εξαιρετικά δεσμενή τα αποτελέσματα και πιο πολύ για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές που είναι πιο τρωτές λόγω των αλλαγών στο κλίμα. Νομίζω πως εκεί είναι τεράστιο το θέμα και πρέπει να το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο πρώτος δωρητής ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και ε, που έχει και τα περισσότερα θαλάσσια σύνορα στον κόσμο. Γι' αυτό θα ήθελα να μας δώσετε μια απάντηση για το τι θα κάνετε. Υποψήφιε Επίτροπος, συμφωνώ απόλυτα πως οι ωκεανοί είναι ουσιαστική σημασίας όχι μόνο γιατί έχω ζήσει στα παράλια σχεδόν όλη μου τη ζωή και γιατί η θάλασσα ήταν τεράστιο κομμάτι της ζωής μου, κυρίως όταν ήμουν πιο μικρή. Έχετε δίκιο λοιπόν, οι ωκεανοί τρέφουν, ε, εξασφαλίζουν διατροφική ασφάλεια, αλλά επίσης και οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουμε πως τα θαλάσσια οικοσυστήματα απειλούνται και αυτό επηρεάζει τη ζωή μας και επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος. Uh, uh, Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, διαθέτει 720 δις ευρώ ε, για το θέμα, οπότε καταλαβαίνετε πως και εγώ θα κάνω ό,τι προσπάθεια μπορώ για να το σπρώξω. Je précise, c'est vrai Τι θα κάνουμε λοιπόν για να αναστρέψουμε αυτή την τάση στα παράλια και στα νησιωτικά και πώς θα επιτρέψουμε στις περιοχές αυτές να ε, ενισχύσουν την οικονομική τους ε, σχέση με τη θάλασσα γιατί ξέρετε πως μέχρι το 2050 το 50% του πληθυσμού θα ζει κάπου κοντά στη θάλασσα και θέλουμε ε, να διατηρηθούν καλύτεροι οι οικογενείς με υγιή οικοσυστήματα γιατί έχουμε τουρισμό, έχουμε διατροφή, παράκτιο πληθυσμού ε, χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για παράδειγμα. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο ε, χρήζει επενδύσεων, ε, έχουμε κάνει αρκετά, αλλά όχι ίσως όσα πρέπει στις παραθαλάσσιες και στις θαλάσσιες περιοχές. Υποψήφια Επίτροπος. Η οικονομική στήριξη προς τους ωκεανούς και η ανάπτυξη αυτών είναι, όπως σας είπα, 720 διορθώνω εκατομμύρια ευρώ, όχι δισεκατομμύρια, και μπορούμε να συζητήσουμε το κατά πόσο επαρκούν ή όχι, αλλά οι ωκεανοί, η αλληλεία θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα του Green Deal, του Πράσινου Συμφώνου. Αυτή ήταν η απάντησή μου και στην κυρία Ριβασί σήμερα. Δεν είναι αρκετό να γίνεται συζήτηση για την εσωτερική διάσταση του Green Deal. Πρέπει να συζητήσουμε και για τις εξωτερικές διαστάσεις του. Και η ωκεανή και αλία θα πρέπει να είναι κομμάτι αυτής της εξωτερικής διάστασης. Έχω την αίσθηση πως έχουμε βρει στήριξη για την ιδέα αυτή, δηλαδή περιβάλλον, κλίμα, να είναι προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον όσο έχει να κάνει με την ε, εργασία των, της, ε, ε, του Κολεγίου των Επιτρόπων. Επόμενος ο ομιλητής, ο Λούις Στέντμαν Μπράις. Εσείς μιλάτε για πάρα πολλά θέματα αναπτυξιακά, αλλά κοιτάξτε κατά τη διαπραγμάτευση του Brexit εσείς ε, μεταχειριστήκατε απέσια και οι συναδελφοί σας το, Ενωμενικό, το Ενωμένο Βασίλειο. Πώς λοιπόν ε, θα έχουμε καλές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες όταν έχετε κάνει προσπάθεια εκφοβισμού ε, ενός ολόκληρου κράτους που ήταν κράτος μέλος. Αυτή τη στιγμή τρέχουν διαπραγματεύσεις για κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο και για τους δύο ο εταίρους. Άρα λοιπόν σε σχέση με τον Brexit θα κάνετε προσπάθειες να αναστρέψετε τις κακές σχέσεις με την προηγούμενη επιτροπή και θα επιτρέψετε ε, να έχουμε μία απλή οικονομική σχέση βιώσιμη μεταξύ μας έτσι ώστε η εταιρική μας σχέση να είναι βιώσιμη. Στο καινούριο σας ρόλο θα επιτρέψετε η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Η υποψήφια επίτροπος. Το Brexit δεν ήταν δική μας απόφαση, ούτε δική μας επιλογή. Όπως και ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος Γιόνκερ έχουν πει στο παρελθόν, λυπάμαι, αλλά σέβομαι το Brexit. Αν επιβεβαιωθεί και υπό την προϋπόθεση πως δεν έχει λάβει χώρα μέχρι τότε το Brexit, θα συνεχίσω να συνεργάζομαι προς μια ε, τακτική αποχώρηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, ρυθμισμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε ε, για το πώς θα γίνει αυτή η αποχώρηση, οπότε δεν είναι σωστό εγώ αυτή τη στιγμή να κάνω οποιαδήποτε δήλωση μελλοντολογώντας για την μελλοντική μας συνεργασία. Αλλά όπως είπα και στην κυρία Μπίλντε, σέβομαι τη δουλειά που κάνει αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο για την αναψυξική συνεργασία και ελπίζω πως ό,τι και να γίνει στο μέλλον θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σχετικά. Επερώτηση. Ο λαός του Ηνωμένου Βασίλειου θέλουν κάποιο είδους απάντηση στα όσα σας ρώτησα. I think we will see that θα δείτε κι εσείς ποια θα είναι η απάντηση και τα αποτελέσματα στο μέλλον. Ας περιμένουμε. Continue with the next question. Επόμενη ερώτηση από τον Κάρλο Σοχίνιο, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Στην επιστολή αρμοδιοτήτων σας ε, αναλάβατε μια συνολική στρατηγική ε, ε, για την Αφρική σε συνεργασία με τον υπατό εκπρόσωπο. Έχουμε και τις διαπραγματεύσεις για μετά το Κοτονού, συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ και την ε, συμμαχία με την Αφρική. Στην επιστολή καθηκόντων σας αναφέρονται οι πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές προτεραιότητες. Δεν αναφέρονται όμως με λεπτομέρεια στο θέμα της βιωσιμότητας. Αλλά η βιώσιμη φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, η επιχειρηματική ελευθερία είναι σημαντικά θέματα. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στην οικονομική και επενδυτική διάσταση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Πώς θα συνεργαστείτε με τον είπατε εκπρόσωπο, ώστε να δώσετε προτεραιότητα στην βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρική σχέση με την Αφρική και τι γίνεται με τον κανονισμό για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και πώς θα φροντίσετε οι εταίροι να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και τα, α, τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και στην Αφρική, οι χώρες εταίροι από την Αφρική. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Η ερώτησή σας πραγματικά είναι κέρια, γιατί Κατά τη γνώμη μου, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση. Όταν μιλούμε για βιώσιμη ανάπτυξη εννοούμε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη. Όλες αυτές οι τρεις πτυχές, η κοινωνική, η οικονομική και η περιβαλλοντική, θα πρέπει να είναι παρούσες γιατί είναι αλληλένδετες και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της ανάπτυξης. Όπως είπα, το πλαίσιο της συνεργασίας μας και ο συνάδελφο το εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιωζέπ Μπορέλ, στενίζεται αυτή την ιδέα. Το πλαίσιο α, της συνεργασίας μας με την Αφρική θα είναι η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πρόγραμμα είμαστε προσιλωμένοι, όχι μόνο εγώ, αλλά το σύνολο ε, των επιδρόπων και φυσικά θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους. Είχαμε την ε, συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στη Νέα Υόρκη και λάβαμε το μήνυμα που είναι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αλλιώς δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030. Οπότε η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η σφαιρική η στρατηγική για την Αφρική είναι ένα ε, μέσο που έχουμε, ένα εργαλείο μας για να αναπτύξουμε εταιρική σχέση με την Αφρική, αλλά και για να υλοποιήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει η στρατηγική όμως να είναι ευρεία, ε, σφαιρική και να περιλαμβάνει τους ε, επιμέρους τομείς. Το εμπόριο, τη γεωργία, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Και ήδη ξεκίνησε συζητήσεις και την προετοιμασία με τον είπατε εκπρόσωπο Ιωζέ Μπορέλ. Πάντως, τονίζω τη σημασία που έχει η προσήλωση του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι μόνο δική μου διαδικασία ή του είπα του εκπροσώπου. Θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα την ασθενίζεται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ για την σαφή απάντησή σας. Όπως ξέρετε, ένα σημαντικό τμήμα της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ είναι ο διάλογος σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανόμενη και της κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Και αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού, έχουμε μια ισομερή κοινοβουλευτική συνέλευση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ, που εξασφαλίζει την κοινοβουλευτική συνεργασία αλλά και την επίβλεψη των προγραμμάτων επιτόπου. Οι χώρες ΑΚΕ έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να παραμείνουν ε, ως ε, ενωμένη ομάδα. Και είπαν στην ε, συνέλευση της ΑΚΕ ότι η νέα συμφωνία μετά το Κοτονού θα πρέπει να περιλαμβάνει μια αντίστοιχη κοινοβουλευτική διάσταση με την προηγούμενη συμφωνία που θα πρέπει να είναι επίσης αυτόνομη. Θα υποστηρίξετε αυτή τη θέση στις, δημογρα... στις ώστε να εξασφαλίσετε τη συνέχεια της ύπαρξης της ομερούς Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και είστε υπέρ αυτής της κοινοβουλευτικής διάστασης και θα την προασπίσετε στις διαπραγματεύσεις. Όπως σας είπα για 16 χρόνια περίπου ήμουν κοινοβουλευτικός ε, και σέβομαι πλήρως το έργο που επιτελείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον είμαι υπέρ της διαφύλαξης της κοινοβουλευτική διάστασης της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δια, αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση. Στα σχέδια που εξετάζουμε υπάρχει η ιδέα τριών περιφερειακών συνελεύσεων στο μέλλον. Όχι μόνο μια ενιαίας ισομερού συνέλευσης, αλλά τριών περιφερειακών συνελεύσεων. Αυτό προβλέπει μέχρι στιγμή στο σχέδιο της νέας συμφωνίας μετά το Κοτονού. Πάντως για μένα το πιο σημαντικό θέμα είναι να μεριμνήσουμε ώστε με τον α ή β τρόπο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να είναι παρούσα η κοινοβουλευτική διάσταση. Αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Και αυτό σίγουρα θα το συζητήσουμε, αν πάρω την εγκρίσή σας φυσικά και αναλάβω τα καθήκοντά μου σε αρχές Νοεμβρίου. Είναι από τις προτεραιότητες μου και η συμμετοχή ε, στην επόμενη κοινοβουλευτική συνέλευση, στην ισομερή συνέλευση, που νομίζω θα γίνει στη Ρουάντα. Η Εύα Κόβατς από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω θερμότατα κύριε Ρουπιλάινεν. Σας ευχαριστώ για τη διεξοδική σας παρουσίαση και εμπεριστατωμένη. Έχω δύο ερωτήσεις το μέχρι τώρα επίπεδο αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας για τις χώρες ΑΚΕ θα διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο υποστήριξης ε, στο επόμενο ΠΔΕΛΤΑΠ για την περίοδο 2021-2027. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιούν ε, αυτά τα σχέδια και προγράμματα θα έχουν την εγγύηση της διατήρησης της χρηματοδότησής τους. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επιτροπέ, έχετε το λόγο. Γνωρίζω ότι η Φιλανδική Προεδρία πραγματοποιεί εργόδης προσπάθειες για την πρόθεση των ε, συζητήσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και όλοι παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις γιατί η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας, η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας φυσικά εξαρτώνται από τη συμφωνία για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων στο ΠΔΠ θα επηρεάσει και τη δική μα χρηματοδότηση, την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Πάντω, προσωπικά με χαροποίησε η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητά αύξηση της χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή συνεργασία. Και Φυσικά θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερους πόρους στην διεθνή μας συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Πριν μίλησα για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Όπως σας είπα, έχω συνεργαστεί με μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη Φιλανδία, οπότε έχω σχετική πείρα και θεωρώ ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι πολύ σημαντικός εταίρος μας και φυσικά θέλω να συνεργαστώ μαζί του στο μέλλον. Επερώτηση από την κυρία Κόπατς. Πολύ σύντομα. Εσείς πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει το Brexit αν συμβεί την αναπτυξιακή και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις χώρες ΑΚΕ. Εσείς πώς αξιολογείτε το πιθανό αντίκτυπο του Brexit αν λάβει χώρα στις εμπορικές ε, σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Υποψήφιο επίτροπος. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερως για το Brexit και όλοι θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στα τέλη Οκτωβρίου. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι δεν είναι δικός μου ρόλος να οικοτολογώ για αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό αργότερα. Μάλιστα. Το, ρόλο, το, το λόγο τώρα έχει συγγνώμη κυρία Μανώ Ομπρή από την ΚΟΕ. Καλημέρα σας. Είμαι απέναντί σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο εκπλήσωμε που δεν έχουμε συζητήσει αρκετά, παρόλο που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Και πρέπει να σας πω πως προχθές εννέα Σουδανοί κατήγγειλαν την BNP Paribas, μια μεγάλη γαλλική τράπεζα, για εγκλήματα πολέμου ε, κατά ε, της ανθρωπότητας και για τη στήριξη του καθεστώτος Αλμπασίρ στο Σουδάν. Με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να λαμβάνουν αποζημιώσεις οι άνθρωποι, γιατί οι πολυεθνικές δρούν ατιμόρυτες. Ε, τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η αναπτυξική βοήθεια περνά όλο και περισσότερο από τη διαδικασία ΣΔΙΤ και πολλές φορές έχουμε και ε, ζώνες ελευθερών συναλλαγών με απόλυτη πρόστασία ε, για τις μεγάλες εταιρείες. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε πραγματική αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να λογοδοτούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, τι θα κάνετε ε, για χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα σύντομα η Γαλλία, η κάτω χώρες ε, για την παρακολούθηση το τι γίνεται στην τροφοδοτική αλυσίδα των μεγάλων επιχειρήσεων. Εσείς θα κάνετε κάτι αντίστοιχο με το, ε, την υποχρέωση επαγρύπνησης όπως κάνει η, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης έτσι ώστε να γνωρίζετε πώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η υποψήφια Επίτροπους. Όπως είπα και προηγουμένως σήμερα και νομίζω ότι αυτή αποτελεί ε, την απάντησή μου στον κύριο Κρέσπο, εμείς θέλουμε ανάπτυξη για τους ανθρώπους. Όχι ανάπτυξη για τις εταιρείε, για τις κυβερνήσεις μας. Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Βέβαια, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως δεν πλήττουμε και δεν βλάπτουμε τους πιο τροτούς, δηλαδή με μείωση ε, της ε, αναπτυξιακής βοήθειας λόγω προβλημάτων της τοπικής κυβερνήσεις. Αλλά κατανοώ πως ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία λύση που θα προσφέρει ωφέλη σε όλους, win-win. Δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο θέλουμε ένα ίσο ε, ίσως κανόνες παιχνιδιούν για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες, μια και διακυβεύονται και οι ευρωπαϊκές θέσει απασχόλησης, αλλά και αυτό που ζητάτε εσείς. Εμείς ως ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προωθούμε ε, τις θέσεις του ΟΗΕ για, τα, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι και η σωστή θέση γιατί όλε οι προσπάθειε που κάνουμε θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη δέσμευση την αναλαμβάνω επερώτηση σε ένα λεπτό. Ξέρετε σίγουρα πως η διαφορά μεταξύ των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών και το αιτήματο δεκάδων ε, μη κυβερνητικών οργάσεων και ε, της κοινωνίας των πολιτών είναι όχι ε, κατευθυντήριες γραμμές αλλά υποχρεωτικές δεσμεύσεις. Υποχρεωτικά στις χώρες αυτές όπου υπάρχει αδύναμο κράτος δικαίου ώστε να λογοδοτούν οι επιχειρήσεις. Υποχρεωτικά. Ναι, να στηρίξουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΕΑ αλλά δεν είναι αρκετό και δεν είναι ο τρόπος να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ΜΚΟ που τους ζητάνε χρόνια. Οπότε θέλω να δω αν μπορείτε εσείς να το δείτε αυτό και να δώσετε κάποια συνέχεια ε, στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν σε μερικές εβδομάδες στον ΟΗΕ για μια ε, παγκόσμια συμφωνία που θα ε, συμπεριλάμβανε κάτι τέτοιο. Ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήταν ιδανικό αυτό για την Ευρώπη. Πείτε μου λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα από μια ανάλυση που έχετε κάνει, ξέρω πώς έχει γίνει και αν θα έχουμε σχέδια εντολή διαπραγμάτευσης ε, έτσι ώστε με ε, στεναρό τρόπο να τα προωθήσει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα σχέση με τις επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποψήφια επίτροπος. Εγώ έχω καταλάβει το εξή. Πρόκειται για μια εντολή για την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, όχι για τη δική μας, γιατί θα γίνει τον Οκτώβριο συνεδρίαση. Αλλά επειδή Έγινε μια ωραία συζήτηση για το θέμα. Έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει ε, μέρος τον Οκτώβριο στη Γενέβη σχετική συζήτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Χρειαζόμαστε να είναι δεσμευτικό το πλαίσιο και θα το μελετήσω, σας υπόσχομαι, πολύ ε, βαθιά το θέμα όταν θα αναλάβω ως Επίτροπος. Τζάκι Jones από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ βρίσκομαι. Κυρία Ουρπιλάινεν, ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας. Για να αναγνωρίσουμε τη δουλειά που κάνουν οι ΜΚΟ επιτόπου και να σας πω τι έχει κάνει ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και επειδή πήρα το προς το τέλος το λόγο και αυτό είναι το καλό. Θα ξεκινήσω με τα εξή. Χαίρομαι για τη δέσμευσή σας ε, για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα ε, ε, των γυναικών, για τις υπηρεσίες αμβλώσεων και αντισύλληψης και χαίρομαι για τη δέσμευση που αναλάβατε για το σχέδιο δράσης για το γένος. Τι θα γίνει όμως με τον προϋπολογισμό, πώς θα εξασφαλίσουμε πως έχουμε κονδύλια επαρκή για μεγάλο διάστημα και πως οι τηρικές αυτές σχέσεις σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών θα ε, ε, συνεργάζονται σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Υποψήφια Επίτροπος, έχω κάτι ακόμα να πω. Η πολιτική συμμετοχή των γυναικών είναι σημαντικό θέμα εμείς είμαστε γυναίκες ε, πολιτικοί και είμαστε παράδειγμα για τις ε, σχέσεις μας ε, με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αν είχαμε περισσότερες γυναίκες πολιτικούς είμαι σίγουρη πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ισότητα των φύλων στις διάφορες πολιτικές. Για την χρηματοδότηση είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που έχουμε ε, επίτροπο για ε, τα θέματα ισότητας των φύλων και με προσδοκία αναμένω τη στενή συνεργασία μαζί της. Νομίζω πως το θέμα είναι τέτοιο που μπορούμε από κοινού να προσφέρουμε έτσι ώστε σε κάθε θέμα πολιτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση του φύλου ε, όσο χρειάζεται. Και αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνει και τη χρηματοδότηση. Δηλαδή να μπορούμε το θέμα αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη στον προϋπολογισμό μας. Είμαι πολύ χαρούμενη ε, για τα όσα θα κάνουμε. Επερώτηση. Είναι καλό που το είπατε, γιατί αυτή η δέσμευση για να στηριχθούν οικονομικά όλες αυτές οι δεσμεύσεις ε, θα ήταν κάτι ακόμα καλύτερο και βέβαια στην ενιαία στρατηγική για την, συγγνώμη, στη σφαιρική στρατηγική για την Αφρική κάτι τέτοιο θα ήταν σωστό, γιατί διαφορετικά για τις ΜΚΟ είναι πολύ δύσκολο και κυρίως λόγω μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται εδώ και 10 χρόνια εκεί το θέμα της χρηματοδότησης έχει ε, πιεστεί και για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρέωσεις μας για την Ατζέντα 2030, όπου είπαμε να μην μείνει κανείς πίσω, θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε και το θέμα της βίας κατά των νεαρών κοριτσιών και είναι σημαντικό όπου και να πάνε να έχουν τη δυνατότητα ε, του να βοηθηθούν όχι μόνο με κονδύλια αλλά και με το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται. Έχουμε και την προτεραιότητα Spotlight που βοηθά νεαρές γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Η υποψήφια Επίτροπος, το ισότητα των φίλων είναι για μένα βασική προτεραιότητα και προσπαθώ πάντα να δοθούν περισσότεροι πόροι στο θέμα. Συμφωνώ μαζί σας, η ισότητα των φίλων χρειάζεται να ε, λαμβάνετε υπόψη σε κάθε είδους ε, πολιτική είναι άλλωστε τμήμα των βιώσιμων ε, στόχων. Ανεπτυξιακών στόχων, τους οποίους έχουμε όλοι δεχτεί. Να σας πω λοιπόν πως εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και την συμμετοχή των γυναικών, χρειάζεται να ακολουθούμε μια τέτοιου είδους ολιστική προσέγγιση και εγώ είμαι έτοιμη να κινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Έλλη από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ως Βρετανίδα ε, Ευρωβουλευτής που πιστεύει ότι είναι σημαντικό προς το δημόσιο συμφέρον να είναι σημαντικός διεθνής εταίρος Ευρωπαϊκή Ένωση και λυπούμε για τη θέση άλλων Βρετανών θα κάνω μια ουσία επί της ουσίας. Για τη ρήπανση και την υγεία θα ήθελα να μιλήσω. Είναι ε, επίσης πτυχές ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, αυτό το τρίπτυχο το, του περιβάλλοντος κοινωνίας και της οικονομίας. Όπως είπατε, το Green Deal είναι προτεραιότητα της εκλεγμένης Προέδρου και σίγουρα είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια. Εσείς μιλήσατε για την εξωτερική διάσταση του Green Deal που δεν φαίνεται μέχρι στιγμής επί χάρτου τουλάχιστον ή δεν προέκυψε στις συζητήσεις. Αυτό με εκπλήσει κάπως γιατί και η ε, έκθεση Lancet ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Υγείας δείχνει ότι η ρήπανση είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό αίτιο της νόσου και των θανάτων γενικώ. Και σκοτώνει τριπλάσιους ανθρώπους από ότι η ελονοσία και η φυματίωση μαζί. Οπότε ε, πώς είναι ε, δυνατόν να αντιμετωπιστεί με λιγότερο ανεπτυγμένα συστήματα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η αναπτυξιακή μας βοήθεια να πιάνει τόπο και να ε, καλύπτει τι ανάγκε κυρίως των φτωχότερων. Είναι διασυνοριακή η ρήπανση του περιβάλλοντος, οπότε τι επιπτώσει τι βιώνουμε όλοι. Ε, θα είστε τμήμα τη ομάδας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μηδενική ρήπανση και θα λάβετε υπόψη αυτή τη προσπάθεια ώστε στην δυνατότητα καταπολέμησης της φτώχειας. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως και είπατε και εσείς, η ρήπανση είναι η σημαντικότερη περιβαλλοντική αιτία για ασθένειες και θάνατο. Και κύριε, δυστυχώς ε, περίπου το 90% των θανάτων αυτών λαμβάνουν χώρα σε ε, χώρες ε, χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Οπότε σίγουρα και το θέμα της ρήπανσης, περιβαλλοντικής ρήπανσης θα πρέπει να ενταχθεί στο πακέτο του Πράσινου Συμφώνου, του Green Deal. Και όπως είπα και νωρίτερα, ελπίζω ότι και εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί και η εξωτερική διάσταση του Green Deal. Και αν συμφωνείτε ως προς αυτό, θα ήταν μια καλή ιδέα να δείξετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υποστήριξή σας προς την ιδέα αυτή γιατί με το Green Deal πιστεύω ότι θα καταφέρουμε ή μπορούμε κατά τη γνώμη μου να στηρίξουμε καθαρή και βιώσιμη ενέργεια για παράδειγμα στις χώρες εταίρους ή να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας ή στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία στις χώρες εταίρους. Οπότε από αυτή την άποψη το Green Deal περιέχει πολλές ευκαιρίες για μας. Και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το, ο Μηχανισμός Γειτονίας Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, το NDICI ή NDICI, είναι σημαντικός. Και με το μηχανισμό αυτό έχουμε με δεσμευτεί να αφιερώσουμε τουλάχιστον 20% ή και περισσότερο στα προγράμματα ε, περιβαλλοντικά ή ε, προγράμματα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και νομίζω ότι είναι πολύ ισχυρή αυτή η και περισσοτερο στα προγραμματα περιβαλλοντικα η ε προγραμματα καταπολεμησης των κλιματικων αλλαγων και νομιζω οτι ειναι πολυ ισχυρη αυτη η δεσμευση μας. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντηση. Είπατε ότι ο τίτλος του χαρτοφυλακίου σας δείχνει ότι θα πρέπει να περάσουμε ε, το, την παλιά διχοτόμηση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αν και θα είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την νέα πραγματικότητα. Ο τρόπο όμω που αξιολογούμε την ανάπτυξη είναι παροχημένο Δεν ε, έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίε. Ε, το ΑΕ κατά κεφαλήν, η ανάπτυξη του ΑΕΠ. Είναι πολύ συσταλτική, περιοριστική η προσέγγιση που έχουμε τη ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη σα πώ θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αξιολογούμε ή που καταμετρούμε την ανάπτυξη, ώστε να λάβουμε υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τη ανάπτυξη, γιατί περιλαμβάνει κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πτυχή. Τι αλλαγέ θα θέλατε, τι δράσει θα αναλάβετε στη διάρκεια τη θητεία σα για να συμβάλλετε σε αυτή την αλλαγή τη ε, προσέγγιση τη ανάπτυξη. Προσωπικά διαπιστώνω ότι αν θέλουμε όντω να υλοποιήσουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που νομίζω είναι κοινή μας επιθυμία, έχουμε ανάγκη μια ολιστική προσέγγιση, μια συνολική σφαιρική προσέγγιση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτή είναι η αναπτυξιακή πολιτική, αυτή είναι η εμπορική πολιτική και αυτή είναι η γεωρική πολιτική και να είναι όλες στεγανά προσδιορισμένες. Αυτά τα στεγανά θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Θέλουμε μια συνολική σφαιρική προσέγγιση που να καλύπτει όλες τις επιμέρους πτυχές. Αν θέλουμε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη ε, και βιώσιμη από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια σφαιρική προσέγγιση ολιστική. Και αυτό είναι ο στόχος της ε, συνολικής μας ε, στρατηγικής για την Αφρική την οποία, επαναλαμβάνω, εστερνίζεται το Σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όλοι συμμετέχουμε στο σχεδιασμό αυτή τη νέα στρατηγική. Όχι μόνο εγώ με τον κύριο Μπορέλ. Και ο Επίτροπο ε, για το Εμπόριο και ο Επίτροπο τη Γεωργία θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτή τη στρατηγική. Και νομίζω αυτό είναι χαρακτηριστικό τη μεταστροφή και της, ε, του περάσματο σε μια νέα προσέγγιση. Αυτή τουλάχιστον είναι η άποψή μου και θα επιχειρήσουμε καλύτερα αποτελέσματα με αυτή τη νέα προσέγγιση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάρτιν Χόργουτ από το Renew Europe. Κυρία Επίτροπε, Δεν θα σας ρωτήσω για τον Brexit και φαντάζομαι να κουφιστήκατε. Ελπίζω πως θα είμαι εδώ και για τα πέντε χρόνια της αιτία μου, συνεργαζόμενος μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τα πολύ δύσκολα θέματα, τα οποία νομίζω χρειάζουν τις προσοχής μας. Τώρα για τη διαφάνεια, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την εισαγωγή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλει το age transparent, η διαφάνεια στην αναπτυξιακή βοήθεια να ενισχυθεί και να πετύχουμε και κάποια πρότυπα διεθνή. Άρα λοιπόν καλό είναι να ξέρουμε πού έχουμε δαπανίσει τα χρήματα που ε, στέλνουμε και επίσης να μειωθεί η ίδια φθορά και να δούμε ε, για ποιο λόγο ε, χρειάζεται η ευρωπαϊκή αναπτυξική βοήθεια και να μην αντιμετωπίζουμε κατηγορίες πως είναι χρήματα τα οποία πηγαίνουν πεταμένα. Άρα λοιπόν τι θα κάνετε για την αύξηση διαφάνειας και τι θα γίνει με τα πρότυπα ΕΑΙΤΕ όχι μόνο μέσα στην ε, Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο ε, πλανήτη. Η υποψήφια επίτροπος. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντική η παρατήρησή σας γιατί είμαι πρώην υπουργό Οικονομικών και γνωρίζω πως πάντα όταν χρησιμοποιεί κανείς τα χρήματα των φορολογούμενων πρέπει να τα χρησιμοποιεί συνετά και με προσοχή και να είναι πάντα κανείς έτοιμος να υπερασπιστεί τον τρόπο με τον οποίο έγινε η χρήση αυτών των χρημάτων. Από αυτή λοιπόν την οπτική γωνία πιστεύω πως χρειάζεται να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, να βελτιωθούμε εκεί. Αν έχετε λοιπόν κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα επίπεδα της διαφάνειας, να σας ακούσουμε. Εγώ είμαι σαφέστατα δεσμευμένη υπέρ της αύξησης διαφάνειας σε οτιδήποτε κάνουμε. Προγραμματισμό, ε, κοινά ε, σχέδια, project. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να εξηγούμε στον κόσμο πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματα αυτά, τι πετύχαμε, ποια είναι τα αποτελέσματα και βέβαια να αποδεικνύουμε πως είμαστε αποτελεσματικοί. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, είναι σημαντικό. Να πω τώρα λοιπόν πως ε, συνεργάζομαι με τη Γενική μου Διεύθυνση εδώ και δύο εβδομάδες και σέβομαι απόλυτα και τις γνώσεις που έχουν και τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, αλλά και την αποτελεσματικότητά τους. Και χαίρομαι που θα έχω αυτή την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί τους και πάλι πιστεύω πως υπάρχει χώρος βελτίωσης. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε κάποιες ιδέες, με μεγάλη χαρά θα σας ακούσω. Ερώτηση. Έχω μια ιδέα. Και είναι σημαντικό να ακούει κανείς ε, τη δέσμευση σε αυτή υπέρ της διαφάνειας. Το χαιρετίζω και είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα του να είμαστε 28 χώρες μαζί. Μπορούμε δηλαδή στα διεθνή βήματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προσωθήσουμε τη διαφάνεια και επίσης τα πρότυπα ΑΙΑΤΗ. Μόνο όμως το ίμιση των κρατών μελών ανταποκρίνονται σε αυτό το πρότυπο. Οπότε είναι δύσκολο για μας να λέμε στον κόσμο ότι εντάξει πρέπει να το σέβεστε κι εσείς όταν μόνο το ίμιση των κρατών μελών το κάνουν. Θα κάνετε λοιπόν προσπάθειες να εξασφαλίσετε στην πενταετή σας θυσία πως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πρότυπο ΙΑΤΗ θα το σέβονται έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη πλατφόρμα για να προωθήσουμε ε, τη ε, διαφάνεια στην αναπτυξιακή βοήθεια παγκοσμίω. Η υποψήφια επίτροπος Είμαι πολύ επιπειραμένη πολιτικός, οπότε ξέρετε προσέχω πάρα πολύ τι υπόσχομαι και υπόσχομαι μόνο αυτά τα οποία μπορώ σίγουρα να τηρήσω. Οπότε δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι θέμα νομιμότητας, νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να είμαστε σε θέση να δείχνουμε στον κόσμο τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε και αυτός είναι ο τρόπος για να ενισχύσουμε και την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα κάνω ό,τι μπορώ. I'll give the Francis Fitzgerald. Francis Fitzgerald. Κυρία Υποψήφια Επιτροπέ, πολύ χαίρομαι που ακούω πώ έχετε αναλάβει, σκοπεύετε να αναλάβετε δράση για την ισότητα των φύλων και το είπατε και σήμερα. Ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουμε ε, του στόχου τη ατζέντα του 2030 και κυρίω του κλιματικού στόχου χωρί σημαντικέ χρηματοοικονομικέ επενδύσει. Η εμπειρία μα από τα μικρά νησιωτικά κράτη δείχνει ότι ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να, να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα στι κλιματικέ αλλαγέ με οικονομική ανάπτυξη και για να μπορούμε και να ανακάμψουμε από ε, φυσικέ καταστροφέ. Πώ μπορεί να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά ε, ιδιαίτερα ευπαθεί περιοχέ και λειτουργώντα και με πολλαπλασιαστικό τρόπο ω προς τη στήριξη άλλων, ώστε να δημιουργήσουμε υποδομέ και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και τις αλλαγέ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και κυρίω για τη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, σημαντικά αυτά που είπατε για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Βεβαίω αυτό θα είναι για μα προτεραιότητα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τι χώρε που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θέλω να τονίσω και μια άλλη πτυχή. Γνωρίζουμε ότι ο ένα και περισσότερε χώρε είναι χώρε μέσου εισοδήματο. Και αυτό είναι κρίσιμη σημασία, διότι αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν διανύσει κάποια απόσταση στην αναπτυξιακή του πορεία. Σε πολλέ χώρε μέσου εισοδήματο οι ανισότητε είναι πολύ έντονες. Υπ' αυτήν την έννοια η προσωπική μου δέσμευση θα είναι να καταπολεμήσω αυτό ακριβώς, τη βάθυνση των ανισοτήτων. Και όχι μόνο στις χώρες μέσου εισοδήματο, αλλά παντού. Σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι μείζον θέμα. Θα είναι λοιπόν αυτό για μένα μια προτεραιότητα, μια κατευθυντήρια γραμμή το πώς θα καταπολεμήσουμε τις ανισότητες με διαφορετικού είδους εργαλεία. Για τον ιδιωτικό τομέα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει ο ιδιωτικός τομέας εδώ να παίξει σημαντικό ρόλο. Με διαφορετικού είδους μέτρα έχουμε το blending, την ανάμειξη εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων και κάποια άλλα. Αλλά στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε μια πλούσια εργαλειοθήκη για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώ αποτελεσματικά τα διαφορετικά εργαλεία. Χωρί όμω τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι μόνο έντιμο και ειλικρινέ να το παραδεχτεί κανεί αυτό. Πρέπει να είναι σοβαρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε κοινού στόχου, οπότε πρέπει να έχουμε και κοινή προσέγγιση. Και αυτό θα είναι μέρο τη δουλειά μα. Επερώτηση. Βεβαίως, Συμφωνώ μαζί σα. Η καταπολέμηση των αξιο... ανισοτήτων πρέπει να γίνει με κάθε εργαλείο που διαθέτουμε. Όμω οι κλιματικέ αλλαγέ δεν είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε καταλήλω και θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερε ανισότητε εφόσον δεν αντιμετωπίζονται. Η ΟΗΕ είπε ότι είναι πολύ απογοητευμένο με το όλο θέμα τη χρηματοδότηση και του πώ διατίθεται για του αναπτυξιακού στόχου και του στόχου τη χιλιετία τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσει συνεργασία μεταξύ δημόσιου ιδιωτικού τομέα, διότι όπως είπα και νωρίτερα, πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις για αυτό το σκέλος είναι πραγματικά πολύ χαμηλές. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι, έτσι είναι για τις κλιματικές αλλαγές. Πολύς λόγος έχει γίνει για, το, για την πράσινη λύση, το Green Deal, είναι ένα παράδειγμα για την ε, δέσμευση τη Μελλοντική Επιτροπή, του Μελλοντικού Κολεγίου των Επιτρόπων και το πώ θα αντιμετωπίσουν τι κλιματικέ αλλαγέ. Η πρωτοβουλία για ένα συνασπισμό όλων των δυνάμεων από τον πρόεδρο Γιούνκερ ήταν μια πολύ καλή ιδέα για να συγκεντρώσουμε και ιδιωτικέ επενδύσει λόγου χάρη για την Αφρική. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Έχουμε ήδη κάποια θετικά παραδείγματα, έχουμε ήδη επιτύχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως υποχρέωσή μου είναι να αναζητήσω νέες πρωτοβουλίες, να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε κι άλλες νέες φρέσκες επενδύσεις στην Αφρική. Είμαι βεβαίως πανέτοιμη να το κάνω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Ναι, Έχουμε ένα δυο λεπτά, αλλά τελείωσε. Περιμένετε, περιμένετε. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Να ευχαριστήσω και την υποψήφια Επίτροπο για όλες τις απαντήσεις της. Σας ευχαριστώ και για τη διάρκεια των απαντήσεων. Φινλανδική αποτελεσματικότητα. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά κανόνες είναι σαφείς. 25 ερωτήσεις. Θα ήθελα πάντως να πω στην υποψήφια επίτροπο ότι εάν επιβεβαιωθείτε και εγκριθείτε, ανυπομονούμε να δούμε πόσο οι δεσμεύσεις που αναλάβατε στις ε, ανακοινώσεις σας και ήταν προσφυλή στο Κοινοβούλιο θα ε, έρθουν και στην, να γίνουν πράξη. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Και καλούμε την υποψήφια επίτροπο αν θέλει να κάνει παρατηρήσεις εν είδη, κάποιες παρατηρήσεις εν είδη συμπεράσματος στην όλη δημόσια κρόαση. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, γιατί μέχρι τώρα δεν την μίλησα σε αυτή την ακρόαση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω δύο κουβέντες στα φιλανδικά. Ευχαριστώ πολύ. Κίτος. Äh, arvoisa Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Όπως επανειλημμένος το είπα από την έναρξη αυτής της ακρόασης, το Ευρωκοινοβούλιο είναι για μένα ένας τόπος σημαντικός. Θεωρώ ότι Εκπροσωπείται πραγματικά την άμεση δημοκρατία και χρειάζομαι και την στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών μέσω ημών των Ευρωβουλευτών για τη μελλοντική μου δουλειά. Ένα μέλλον αηφόρο βιώσιμο είναι εφικτό μόνο εφόσον υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που μου φέρατε αυτές τις ερωτήσεις εν είδη προκλήσεων για να μπω στην ουσία του θέματος, στην ουσία των αρμοδιοτήτων μου. Η ακρόαση αυτή αντικατοπτρίζει την μεγάλη σημασία αυτού του τομέα. Θα ήταν σημαντικό τις εταιρικέ σχέσεις να τις ε, σχεδιάσουμε μαζί, σε συνεργασία με σας. Η όλη συζήτηση κατά την άποψή μου εκφράζει την εκτίμησή μας και την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει η αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι πραγματικά στο επίκεντρο της προσοχής. Όταν το Ευρωκοινοβούλιο ε, πρόκειται να αφήσει το αποτύπωμά του, το, τα ίχνη του, τι ζωέ, τι συνθήκε διαβίωσης δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον ε, κόσμο. Αυτό Το χαρτοφυλάκιο επίσης, έτσι όπως θα είναι ανανεωμένο, θα βρίσκει και στην πρώτη γραμμή της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντικατοπτρίζει την πολύτιμη παράδοση που ε- ήδη έχουμε καταρτήσει σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασία, αλλά και κάτι ακόμα, ότι έχουμε ακόμα κάποιες ευκαιρίε για να εκφράσουμε το λόγο, την άποψή μα και να επηρεάσουμε την ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο, σε ισότιμοι εταίροι με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε συνεργασία. Η εξάλληψη της φτώχειας είναι στο επίκεντρο της δουλειάς μας. Πρέπει να ανακόψουμε την άνοδο της φτώχειας παντού Έχουμε μπόλικη δουλειά μπροστά μας, διότι ακόμη 70 εκατομμύρια πολίτες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να φτάσουμε το στόχο του 0,7% επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στα πλαίσια της πολιτικής μας. Πρέπει να έχουμε πραγματικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ ισοτήμων εταίρων. Δεν μπορούμε μονομερώς να προσφέρουμε βοήθεια ως ελεημοσύνη. Πρέπει να ε, αντιμετωπίζουμε από κοινού τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε τις δομές διαλόγου που έχουμε αναπτύξει με τους εταίρους μας και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης δείχνουν ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στον 21ο αιώνα. Αυτοί οι 17 στόχοι μας δείχνουν ακριβώς ποιος είναι ο προορισμός μας, ποιος θα έπρεπε να είναι ο προορισμός μας. Και αν συγκρίνουμε αυτού του στόχου με το τι συνέβαινε παραδοσιακά στην αναπτυξική βοήθεια, φαίνεται ότι χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου, περισσότερα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια. Χρειαζόμαστε με κυβερνητικέ οργανώσει και ιδιωτικέ εταιρείε να είναι δεμένε στο άρμα αυτό των στόχων τη αναπτυξιακή πολιτική. Και θα πρέπει επίσης τα πρότυπα και οι αξίες μας να λαμβάνονται υπόψη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επενδύσει δημιουργούν θέσεις εργασίας για αυτούς που δεν τις έχουν. Είμαι πεπισμένη ότι αυτές οι εταιρικέ σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο θα μου επιτρέψουν και μένα στη δουλειά μου να επικεντρωθώ στην επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, στην εκρίζωση των ανισοτήτων και την εξάλληψη της φτώχειας. Αυτό είναι το πεδίο εντός του οποίου θέλουμε να κινηθούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας για παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη. Φίλοι μου, είμαι εκφύσεως αισιόδοξη συμφωνώ με τον Μαχάτ Μαγκάντι στο αξίωμά του ότι η ανθρώπινη ζωή είναι σαν ωκεανός. Μπορεί να υπάρξουν και φορτούνες στον ωκεανό ή κυλίδες ρήπανσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ωκεανός είναι όλος μολυσμένος. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικέ γενιές. Και πραγματικά να ολοκληρώσω λέγοντα ότι είμαι υπερήφανη για μα και την Ευρώπη. Η συζήτησή μα δείχνει για άλλη μια φορά ότι η κοινή μα δουλειά επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουμε πρωταγωνιστή στα διεθνή πράγματα. Και έτσι θα πρέπει να μείνουν τα πράγματα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. And on that note, we end this public hearing. Και λύεται η συνεδρίαση και ολοκληρώνεται η δημόσια κρόση.